Καλώς ήρθατε κύριε Ποτόσνικ. Θα ξεκινήσουμε τώρα με την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης. Παρουσίαση που θα μας κάνει ο Διευθυντής του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας, ο κύριος και ο κύριος Ροτμόν που είναι πρόεδρος της ΣΑΡ. Έχουμε στη διάθεσή μας μία ώρα, 60 λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με ένα 20 λεπτό για τους ομιλητές μας. μπορούν να μιλήσουν όπως τους αρέσει και μετά θα έχουμε συζήτηση με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας, ε, κυρία Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας κάνω αυτή την παρουσίαση. Το έγγραφο μοιράζεται αυτή τη στιγμή, είναι οι διαφάνειες που έχουμε φτιάξει. Δεν θέλουμε να τις δούμε μία-μία ξεχωριστά όμως μπορεί να σας χρησιμεύσουν γιατί μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που ίσως έχετε και γι' αυτό μπορεί να κάνουμε κάποιες παραπομπές και μία αναφορά στις διάφορες διαφάνειες που απαρτίζουν το έγγραφο που σας έχει μοιραστεί. Έχουμε όμως μία κύρια διαφάνεια την οποία θα προβάλλουμε στην οθόνη. Είναι η παρουσίαση της ε, δεύτερης έκθεσης παρακολούθησης ε, της αγοράς που συντάσσεται σε αιτήσια βάση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού ε, αερίου. Και καλύπτουμε τρεις τομείς, ε, τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, την αγορά φυσικού αερίου και την αγορά λιανικής. Ασχολούμαστε με θέματα προστασίας του καταναλωτή και απόκτησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την αγορά χονδρικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είδαμε τις εξελίξεις στην αγορά χονδρικής το 2012 και εδώ έχουμε τις συστάσεις και τα συμπεράσματα. Και αυτά βασίζονται στις αναλύσεις και θα έχετε την έκθεση αύριο η σύζευξη, η τιμολογιακή, η σύνδεση της τιμής είναι αυτό που οδηγεί τις τιμές να συγκλίνουν και την αγορά να γίνεται όλο και πιο ολοκληρωμένη. Έχουμε αποτελεσματική χρήση της διασύνδεσης. Εάν δείτε τη διαφάνεια υπαριθμών 14, θα δείτε ότι στην περίοδο μετά το 2008 αυξήθηκε η σύγκληση των τιμών σε πολλές περιφέρειες στην Ευρώπη. Δηλαδή οι τιμές άρχισαν να εξελίσσονται αρκετά, με αρκετά παρεμφερή τρόπο, τρόπο ε, στους, στις ίδιες περιοχές σε όλη την περιφέρεια εκτός από την περσινή χρονιά και σε αυτήν θα επανέλθω. Αυτό οφείλεται στη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στο φαινόμενο των look flows. Το μήνυμα που έχουμε αποκομίσει είναι το εξή. Η πλήρη υλοποίηση του μοντέλου μας πρέπει να είναι προτεραιότητα, να παραμείνει προτεραιότητα αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει διαχείριση για την αποσυμφόρηση, αυτό να εγκριθεί τάχιστα και να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν ε, ταχύτερα οι διατάξεις. Αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για σήμερα και για το μέλλον. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς μέχρι το 2015. Και αν δείτε τη διαφάνεια 16, τότε θα αντιληφθείτε ότι είναι πολλά τα ωφέλη της ολοκλήρωσης ή της αγοράς, της ε, φυσικής σύνδεσης αν θέλετε μεταξύ των κρατών μελών. Και θα δείτε τι, ποιο είναι το διακύβευμα από πλευρά ωφελιών για τον τελικό καταναλωτή. Θα πρέπει η σύζευξη αυτή να παραταθεί, να επεκταθεί πέραν της υφιστάμενης κατάστασης. Δηλαδή Θέλουμε μέχρι τα τέλη της επόμενης χρονιάς, ε, σε όσο περισσότερες περιοχές στην Ευρώπη, να έχουμε αυτό το market coupling. Δυστυχώς ε, τα πράγματα δεν πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση σε πολλές περιπτώσεις φαίνονται αυτές στη διαφάνεια υπαριθμών 15 ως προς την ηλεκτρική ενέργεια. Στην νοτιοδυτική Ευρώπη ισχύει αυτό. Εδώ έχουμε σύζευξη στην αγορά σε μεγάλο βαθμό. Αυτό ισχύει για τα περισσότερα σύνορα στην περιοχή και το επίπεδο των ροών που αντίκεινται ε, στο, στην κατεύθυνση του διαφορικού τιμής έχει πέσει στο μηδέν. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να επιτύχουμε σε όλη την Ευρώπη. Ελπίζουμε μέσα σε ένα μισή χρόνο και καλύτερα θα ήταν να τα πετύχουμε νωρίτερα. Ε, η, η δυνατότητα του συστήματος δεν περιορίζει την ολοκλήρωση της ε, ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη. Αυτό το βλέπετε και στα δεξιά στη διαφάνεια υπαριθμών 15. Και θα πρέπει επιγόντως να ρυθμίσουμε ε, το θέμα των μη προγραμματισμένων ε, κενών ε, στην ροή, των μη προγραμματισμένων ροών. Έχουμε τη σύγκληση τιμών το 2012, αυτό αυξήθηκε σε πολλές περιοχές και αυτό εν μέλει οφείλεται σε, σε αυτά τα loop flows. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε και να βρούμε λύση τόσο βαραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη. Και τέλος, θα αποκομίσουμε μεγάλο όφελος από το να ε, ε, εξελιχθούν με, με συνέπεια η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η αγορά φυσικού αερίου εάν έχουμε μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στρέφομαι τώρα στις αγορές φυσικού αερίου. Έχουμε απώλειες για τον Ευρωπαίο καταναλωτή, συνεχίζονται αυτές, διότι δεν υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Είναι κατακαιρματισμένη η αγορά και δεν υπάρχει απόλυτη ολοκλήρωση. Σαφέστατα λοιπόν σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση το, τα επόμενα χρόνια. Να υλοποιήσουμε τη διαδικασία διαχείρισης της αποσυμφόρησης και της συμφόρησης capacity congestion procedure mechanism και θα πρέπει να επιταχύνουμε την ε, ε, εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Ακόμα ε, και, αν δεν γίνουν, ακόμα και πριν να γίνουν νομικώς δεσμευτικά αυτά τα κείμενα. Στη διαφάνεια 24 βλέπετε ότι έναντι υψηλού επίπεδου ε, κλεισίματος ε, ε, μακροπρόθεσμου της δυναμικότητας διασύνδεσης από τη μία χώρα στην άλλη. Έχουμε χωρητικότητα και δυναμικότητα η οποία την κλείνουμε την ενσωματώνουμε μακροπρόθεσμα, αλλά τελικά δεν τη χρησιμοποιούμε στην πράξη και παραμένει ε, ως ίζημα, αν θέλετε, παραμένει αδρανής. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η χωρητικότητα να ξαναμπεί στην αγορά. Και θα πρέπει να προωθήσουμε τη σύγκληση των μακροπρόθεσμων συμβολέων και των ε, ε, συναλλαγών ε, on the spot. Στη διαφάνεια επαριθμών 20 βλέπουμε το γεγονός ότι οι τιμές εξέλιξης Ε, ταυτίζονται με καθυστερήσεις. Δεν έχουμε πετύχει την αποσύνδεση των τιμών συμβολέων φυσικού αερίου ε, μεταξύ αυτών και των ε, άλλων τιμών. Και επομένως οι τιμές του φυσικού αερίου δεν αντικατοπτρίζουν τις βραχυπρόθεσμες συνθήκες στην αγορά και άρα δεν υπάρχει κίνητρο το φυσικό αέριο να κυκλοφορήσει ευρύτερα στην Ευρώπη. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε κανόνες για hub trading, για να έχουμε περιφέρειες που θα εμπορεύονται και θα γίνεται εκεί το, οι συναλλαγές θα γίνονται και να βελτιώσουμε την εναρμόνιση των ε, διασυνοριακών δασμών μετάδοσης και μεταφοράς. Στο διαφάνεια 32 βλέπετε πως έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή και θα δείτε ότι είναι τεράστια διαφορά μεταξύ ε, της τιμής, της ταρίφας, όχι δασμού, με συγχωρείτε, ε, transmission, από τις ίδιες χώρες και από πλευράς φυσικού αερίου θα υπάρξουν και ωφέλη για περαιτέρω ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου γιατί η αγορά φυσικού αερίου μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα παραγωγής και προμήθευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. <coughs> να στρεφώ τώρα στις αγορές λιανικής. Δυστυχώς Ακόμη βρίσκουμε να υπάρχουν ε, χαμηλά ποσοστά στα, χαμηλές, χαμηλή επιτυχία στα ποσοστά μετατροπής στα κράτη-μέλη. Και αυτό διότι υπάρχει η προσκόλληση στους ε, τοπικούς ε, παρόχους του μεθευτές και οι δραστηριότητε αυτές κάποιες φορές φαίνονται περίπλοκες, χρονοβόρες και ρηψοκίνδυνες. Ξέρουμε ότι 23 μάλλον για 23 χώρες για την ηλεκτρική ενέργεια και για, τις 18, ε, για το, και για 18 για το φυσικό αέριο καταφέραν να κάνουν κάποια μετατροπή, αλλά η ρύθμιση των τιμών παρέμεινε πρόβλημα. Είναι δύσκολο να έχουμε σύγκληση 49% για την ηλεκτρική ενέργεια και 46% για το φυσικό αέριο από το μερίδιο της αγοράς δεν έχουν ρυθμισμένες τιμές. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την μετατροπή οι καταναλωτές και το τελικό κόστος ε, είναι υψηλό, γι' αυτό είναι ένας φραγμός στο να το επιλέξουν. Ως προς τα ρυθμιστικά εμπόδια υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά καθεστώτα και διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα τα οποία δημιουργούν ε, περιπλοκότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την αδειοδότηση. Είναι διαφορετικό το σύστημα μεταξύ των κρατών μελών. Η πλήρης αποσύνδεση πάντως δεν έχει επιτευχθεί και σε πολλά κράτη δεν εφαρμόζεται καν. Και αυτό έχει να κάνει πολλές φορές και με την νέα επωνυμία που πρέπει να λάβουν οι προμηθευτές της Λιανικής. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που οι τιμές της Λιανικής αυξήθηκαν ε, φέτος και υπονολογίζεται να συμβεί και του χρόνου, παρά την οικονομική ύφεση. Ενώ έχει μείνει σταθερή η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι φόροι και οι δασμοί σε κάποια κράτη-μέλη έχουν περιορίσει την ε, προσαρμογή της τιμής σε ένα 50%. Και σε πολλά κράτη-μέλη παραμένει μια βασική ανησυχία το θέμα της προμήθειας της τροφοδότησης σε ενέργεια. Θα πρέπει μάλιστα να γίνει κάτι και για να καθησυχαστούν οι καταναλωτές αλλά και να ρυθμιστεί σωστά η ανταγωνιστικότητα. Για τις τιμές θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το κόστος εισόδου ώστε να, υπάρχει, να υπάρχουν σωστή όροι ανταγωνισμού. Και οι τιμές θα πρέπει να σταματήσουν να πιέζονται ώστε να μπορέσουν και τα υπόλοιπα κάτι μέλη να είναι ανταγωνιστικά. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να δερματίζουν ενεργό ρόλο ώστε να εφαρμοστούν τα μέτρα του τρίτου πακέτου και να λάβουν πια και οι καταναλωτές τα ωφέλη από την μετατροπή, αλλά να ενισχυθούν και τα δικαιώματά τους. Μερικά συμπεράσματα για τις ανισότητες και για το πώς ε, τα μέτρα που αφορούν τους καταναλωτές από το τρίτο πακέτο είναι υπόθεση των κρατών μελών που θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι ορισμοί είναι ένα θέμα, όπως για τον ευάλωτο χαρακτήρα ή το τι γίνεται με την περίπτωση της πτώχευσης. Δεν έχουν όλα συγκεκριμένο ορισμό για το τι είναι ένας ευάλωτος καταναλωτής και τα μέτρα για να προστατευτούν αυτοί οι καταναλωτέ ε, διαφέρουν. Διαφέρουν μέσω τη νομοθεσία για την πρόνοια ή για την ενέργεια ή ένα συνδυασμό και των δύο. Το επίπεδο συμμόρφωση με, την ενημέρωση, με τι απαιτήσει για ενημέρωση του καταναλωτή από το τρίτο πακέτο είναι αρκετά υψηλό και αυτό το σημειώνουμε με ικανοποίηση στα περισσότερα κράτη-μέλη. Οι περισσότεροι έχουν ανεξάρτητο φορέα επίλυση διαφορών 20 ε, για το αέριο και 25 για την ηλεκτρική ενέργεια. Κάποιες φορές μιλάμε για γενικές ή ειδικέ ε, φορείς που ασχολούνται γενικώ ή ειδικώ με την παροχή ενέργειας. Επίσης ε, συλλέγονται δεδομένα για όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε διαφορετικό βαθμό μεταξύ των κατών μελών, οπότε θα πρέπει να υπάρξει ε, καλύτερη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων σε σχέση με, την, με τις προσφυγές, τις διαφορές. για την ευφυή μέτρηση Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ κρατών μελών. Κάποιοι 20 έχουν μέτρα για την περίπτωση του αερίου και 24 για την ηλεκτρική ενέργεια. Και εδώ χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω βελτίωση. Σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα, τα συμπεράσματα για το τι συμβαίνει, παρά την οικονομική ύφεση της τελευταίας διετίας, ε, τα νοικοκυριά της Ευρώπης ε, ουσιαστικά πρέπει να υποστούν τις αυξημένες τιμές. Ε, το γνωρίζουν οι συνάδελφοι, είναι κάτι που διαρκώς αυξάνεται. Αλλά ενώ βελτιώνεται η κατάσταση της αγοράς, η συμπερίληψη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα διάφορα κενά που παραμένουν εμποδίζουν τη σύγκληση των τιμών. Και αυτό γιατί δεν είναι διαφανές το σύστημα της ε, φορολόγησης της μεταφοράς αερίου. Η ανταγωνιστικότητα στις αγορές των περισσότερων κρατών μελών τονώνεται, αλλά πρόοδος χρειάζεται περαιτέρω. Η μετατροπή δεν είναι ακόμη επαρκής. Οι τιμές δεν είναι ακόμα ρυθμισμένες πλήρως μεταξύ των κρατών μελών, οπότε αυτό δεν δημιουργεί εμπιστοσύνη στους καταναλωτές. Παραμένουν μεγάλα ζητήματα αυτά. Τέλος, οι βασικές μας ε, συστάσεις. Δεν είναι περίεργο που απαιτείται πλήρης εφαρμογή, πλήρης υλοποίηση του τρίτου πακέτου όπως πολλές φορές έχει πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί όχι μόνο από την Επιτροπή που θα πρέπει να πιέσει με τη σειρά της τα κράτη-μέλη, αλλά και με τις ρυθμιστικές αρχές των ε, κρατών μελών που θα πρέπει και αυτές να εργαστούν. Η εφαρμογή του κανόνων για το πρώτο δίκτυο, για το, για το πρωτογενές δίκτυο, είναι ήδη κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα ενώ η επίλυση των ε, διαφορών, η αντιμετώπιση των προσφυγών και το τι γίνεται με τα κενά και τις ελλείψεις που παραμένουν από πολιτικής, χρήση πολιτικής δράσης. Επίσης για, τις, για τους δασμούς μεταφοράς και την ε, περίπτωση του υγροποιημένου αερίου πρέπει να επιδείξουμε περισσότερη διαφάνεια, ώστε οι καταναλωτές να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να μπορέσουν να ωφεληθούν από τη μετατροπή για να έχουμε μια ανταγωνιστική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει πλήρης εφαρμογή και των δικαιωμάτων που μπορούν να ασκήσουν οι καταναλωτές. Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν για αυτό το πολύ χρήσιμο κείμενο, νομίζω 270 σελίδες, μακροσκελέστατο έγγραφο, με πάρα πολλές πληροφορίες και κατά δεύτερον αυτή είναι η κατάσταση στη σημερινή φάση. Όμως έχουν αρχίσει διαβουλεύσεις, μάλλον προετοιμασία για διαβουλεύσεις, οπότε ευχαρίστω να παράσχουμε πληροφορίες για αυτό που έχουμε ονομάσει Πασαρέλα για το 2025. Ε, ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει η μετάβαση προς τα μέσα της δεκαετίας του 2020 να γίνει ομαλός, χωρίς να επικεντρωθεί μόνο στο άμεσο παρόν. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι και η έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στη σημερινή συζήτηση. Bene, voi avete terminato. Bene, allora alla fine... Μετά τις ε, παρουσιάσεις αυτές, ο πρώτος εγγεγραμμένος αγορητής είναι ο συνάδελφος Τούρμες. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Έχω ένα ερώτημα στο θέμα της υλοποίησης. Ήταν μία απέτηση κλειδί στην έκθεση του κυρίου Μπούζεκ και ρωτώ την Κομισιόν σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στον προγραμματισμό δεδομένου ότι ορισμένοι κωδικοί είναι έτοιμοι να αποφασιστούν. Πότε θα μπορέσει αυτή η τελική φάση να περάσει από την επιτροπολογία και εν συνεχεία θα γίνει επιτροπολογία με ενδελεχή μελέτη ε, ή πώς θα επιταχύνουν τη διαδικασία για να μην σταματήσουν οι διαδικασίες από τον Απρίλιο και πέρα και να τελματώσουν τα, τα πράγματα. Ε, το ουσιαστικό πρόβλημα της Ευρώπης όσον αφορά την τιμολόγηση είναι το φυσικό αέριο. Και κάναμε μια πολύ έντονη έκκληση και στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και σε όλους τους συναρμόδιους να σταματήσει επιτέλους αυτή την ε, ιστορική, τον ιστορικό αναχρονισμό της φορολόγηση των ε, τιμών του πετρελαίου. Διότι η φορολόγηση μας επιβαρύνει πολύ περισσότερο το πετρέλαιο από ό,τι στην Αμερική. Πρέπει λοιπόν να ε, βοηθήσουμε τον ανταγωνισμό και πρέπει να μας πείτε εσείς τι μπορούμε να κάνουμε εμείς περισσότερο από αυτή τον πόλεμο που κάνει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στην Gazprom. Τρίτον, ευχαριστώ τα σχόλιά σας για τη, στη σελίδα 17 για το κλείσιμο του, του loop, του, του κόμβου. Διότι οι μεγαλύτερες ε, πηγές ε, το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος κόμβος nuclear exports. That's because, that's why Slovenia... Α, ε, είναι 500 από τη Γερμανία στην Πολωνία, δεν περνάει, αλλά αυτό το, το loop ε, τότε πρέπει, που λέτε ότι πρέπει να κλείσει πρέπει να ε, αναφέρεστε στην ε, πυρηνική ενέργεια. Εάν λοιπόν εσείς αντί για την πυρηνική αναφέρεστε στην αιωλική ενέργεια, τότε έχουμε πρόβλημα, διότι αυτή η κομβική σχέση δεν περνά διασυνοριακά και χρειάζεται να δράσουμε. Όταν ε, κάναμε τη δεύτερη μελέτη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ε, κάναμε τεράστια μάχη για να πείσουμε τους καταναλωτές να αλλάξουν. Προμηθευτή, προμηθευτή. Και η Άντζελα, ε, όχι Άντζελα γιατί είναι κάποια άλλη κυρία που ανακατεύεται στη γερμανική πολιτική, η Αντζέλικα μετά από ε, ένα πυροβολισμό ε, ε, ειδήσεων προς τον καταναλωτή ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπερβολικά υψηλό και δεδομένου ότι η Γερμανία ενημερώνει τους καταναλωτές μέσω του διαδικτύου και της ενημέρωσης. Αφού βομβαρδίσαμε λοιπόν τους καταναλωτές πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να τα κορουθεί όλα αυτά σαν να είναι η καθημερινή του εργασία. Και αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή εσείς χάνετε, ε, έχετε χάσει από τα, μάτια, μάτια σας, είναι ότι ε, ο καταναλωτής δεν μπορεί να παρακολουθήσει πια την τιμολόγηση και στη Λιψία έχει κατεβεί σημαντικά το κόστος της ε, κιλοβατόρας ε, στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντικά ε, στο μεγαλύτερο, στη μεγαλύτερη μονάδα που βρίσκεται στη Λιψία. Παρόλο λοιπόν που έχει κατεβεί το κόστος παραγωγής και διανομής, ο Γερμανός καταναλωτής δεν έχει υποφεληθεί ούτε ένα σέντς. Και ερωτώ, Πού διαφεύγει όλο αυτό το χρήμα που εξοικονομείται. χρημα που εξοικονομειτε εσεις μας είπατε ότι η αγορά spot δεν είναι η αγορά future, αλλά εν πάση περιπτώσει μετά από 3-4 χρόνια μειώσεως του κόστους δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο η τιμή χρέωσης στους καταναλωτές δεν μπορεί να κατέβει. Είναι μια, ε, μια ανομαλία της αγοράς η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί περαιτέρω, είναι απαράδεκτη ε, και θέλω να ξέρω σε πού οφείλεται αυτή η ακαμψία και η μη μείωση του, της τιμολόγησης. Ευχαριστούμε κύριε Τούρμες, ο κύριος ε, Είχα την εντύπωση ο κύριος Τούρμες μίλησε τόσο ωραία για αυτή την δυναμική γυναίκα που αναφέρθηκε ε, που θα ήθελα να τον ακούσω και λίγο παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, σας συγχαίρω για την εισήγησή σας και την έξεση σας και πολύ χαίρομαι που δεν μας την παρουσιάζετε σελίδα προς σελίδα, τόσο μεγάλη που είναι. Και θέλω να ρωτήσω πώς θα αντιμετωπίσετε τις ε, πολιτικές ε, πτυχές, την πολιτική και καταναλωτική αντίδραση στις αυξανόμενες τιμές. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο πολύ μπερδεύει τους καταναλωτές γιατί βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν, οι χρεώσεις να ανεβαίνουν τη στιγμή που η ευρωπαϊκή οικονομία είναι πιεσμένη θα έλεγα και όχι τελείως συμπιεσμένη. Τέλο πάντων δεν λειτουργεί με πλήρες ε, δυναμικό. Ε, και Έχουμε μια κατάσταση που οι, τα ορυκτά, οι πηγές ε, ενέργειας είναι επαρκέστατες και όμως υπάρχει μια απόλυτη αποσύνδεση μεταξύ αυτών των πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου. Δεν βλέπω πώς θα συνεχιστεί αυτή η ανομαλία. Είναι μεγάλο πολιτικό το θέμα, διότι βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο σε μια κατάσταση στάσιμων εισοδημάτων, εν ώψη μιας ενεργειακής κρίσης, όχι μόνο έρχεται, και οι καταναλωτέ ε, πιστεύουν ότι είναι υποχρεωμένοι να μειώσουν την κατανάλωσή τους γιατί δεν μπορούν να, την να πληρώσουν το κόστος. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, την ε, φύλαξη ε, του Κλόντ για την αλλαγή προμηθευτών, ε, των παρόχων μάλλον ενέργειας, δεν λειτουργεί, δεν δουλεύει το σύστημα. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ full time με το ποιος είναι ο καλύτερος πάροχος και να αρχίσω να ψάχνω και το ηλεκτρικό και τους παρόχους φυσικού αερίου, ποιος είναι ο καλύτερος, να παίρνω τηλέφωνο, να ψάχνω τα τιμολόγια ε, δεν, ε, δεν μπορεί να δουλέψει αυτό το σύστημα στο επίπεδο που το θέλουμε εμείς και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να ενσαρρύνουμε τους καταναλωτές. Βεβαίω ο ανταγωνισμό είναι ένα από του τρόπου με του οποίου μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό ε, των τιμών. Αλλά ο Κλοντ και <laughs> είναι αντιπωσιακό αλλά φαίνεται ότι συμφωνώ εδώ μαζί του. Ε, τι θα κάνουμε έναντι του καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν πρέπει να το κάνουμε τη ζωή πολύ πιο δύσκολη, αλλά πιο εύκολη. Εγώ έχω πίστη στις ρυθμιστικές αρχές, δηλαδή η εμπιστοσύνη ότι μπορούν να πράξουν, να ενεργήσουν. Τι θα πούμε λοιπόν στους καταναλωτές μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντλήσουν ε, κάποια αισιόδοξα μηνύματα για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε ε, την αγορά του της ε, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή είμαστε ακόμα κολλημένοι στο πρόβλημα της Gazprom. Ευχαριστούμε. Ο λόγος του συνάδελφου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που έχουμε σήμερα την ε, ευκαιρία να κουβεντιάσουμε περισσότερο για την κατάσταση της αγοράς ενέργειας ιδίω για την εσωτερική αγορά της Ευρώπης στην ενέργεια. Καλώς ορίζω τον κύριο Ποτόσνικ, τον διευθυντή της ε, Acer που έχει και την έδρα της στην Σλοβενία. Έχω δύο ερωτήσεις, εάν με επιτρέπετε. Πρώτον, έχω πολλά στοιχεία από την τελευταία διετία ότι στην Acer υπάρχει έλλειψη πόρων, έλλειψη κονδυλίων. Και αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Είναι όλα εντάξει πλέον ή υπάρχουν ακόμη εκκρεμή ζητήματα σχετικά. Και το δεύτερο. Η Acer είναι στη Σλοβενία όμως η Σλοβενία αυτή τη στιγμή έχει από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, χονδρικός. Εδώ λοιπόν αναρωτιέμαι τι συμβαίνει και είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Ευχαριστούμε ο συνάδελφος Κρόλη. Ευχαριστώ. Τρία είναι αυτά που μου τραβούν την προσοχή ως προς τις παρουσιάσεις που ακούσαμε σήμερα. Πρώτον, οι τιμές ε, του ηλεκτρισμού ανέβηκαν και για τους καταναλωτές και στη βιομηχανία. Οι τιμές του φυσικού αερίου επίσης ανέβηκαν και για τους βιομηχανικούς χρήστες και για τους καταναλωτές, τους ιδιώτες. Και όταν μιλούμε για την αλλαγή, το να πάει κανείς από ένα πάροχο υπηρεσία σε κάποιον άλλον, αν το έχει αν το έχετε κάνει ποτέ, το έχετε δοκιμάσει, σας παρουσιάζουν διάφορες τιμές τις οποίες για να καταλάβετε πρέπει να είστε και μηχανολόγος και μαθηματικός, για να καταλάβετε ποιο σας συμφέρει περισσότερο. Και η δυσκολία να αλλάξει τελικά κανείς πάροχο και γι' αυτό κάνουμε και μακροχρόνιες συμβάσεις ω καταναλωτές, είναι και το μεγαλύτερο αντικίνητρο. Αντικίνητρο και γι' αυτό ο κόσμος δεν ψάχνει ένα καλύτερο deal, μια καλύτερη προσφορά για να πέσουν τελικά οι τιμές. Και οι ιδιώτες είναι και οι πιο ευαίσθητοι, αν θέλετε, χρήστες που πλήττονται περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι πλήττονται περισσότερο όσοι είναι στις παρυφές, όσοι έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα ανεξαρτήτως ε, διάρθρωσης ε, της φορολογίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Και παρόλο που Έχουμε αυτό το ιδανικό της μίας ενιαίας αγοράς ενέργειας και στην παροχή της, στην προμήθευσή της αλλά και στη χρήση της τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι και στις δικές σας διαφάνειες φαίνεται ότι υπάρχει τεράστια διασύνδεση και διαθεσιμότητα εναλλακτικού παρόχου στην κεντρική Γαλλία, από τη Γερμανία στην Πολωνία, από το Βέλγιο στις κατοχώρες, από τη Γαλλία στην Ιταλία αν θέλετε, αλλά όσο πιο απομακρύνεται κανείς από το κέντρο, τόσο πιο δύσκολο είναι εκεί να γίνει αυτό το πράγμα. Σουηδία, Φιλανδία, μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, Ιρλανδία, χώρες της Βαλτικής δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορούν να έχουν τόσες πολλές εναλλακτικέ πηγές αυτές οι χώρες και εναλλακτικού παρόχους και εναλλακτική προμήθευση σε οτιδήποτε. Μπορεί να μην έχει άμεση σχέση αυτό που λέω, αλλά το συζητήσαμε και με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν συζητούσαμε για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τους ε, interconnectors. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε εναλλακτικού παρόχους, και για να είναι βιώσιμοι σε αυτές τις χώρες που ουσιαστικά είναι απαγορευτική η ύπαρξή τους, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα, να υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες για αυτούς. Στο BBC News είδα χθε βράδυ ότι τα κέρδη των έξι μεγαλύτερων εταιριών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέβηκαν από 340 εκατομμύρια στερλίνες το 2006 σε 1,1 δις στερλίνες το 2012 ενώ όλες οι άλλες τιμές πέφτουν και της ακίνητης περιουσίας και των βασικών αγαθών και οποιοδήποτε άλλου προϊόντος. Κάθε φορά λοιπόν που πέφτουν οι τιμές, τεράστια κέρδη αποκομίζει η εφοδιαστική αλυσίδα, η αλυσίδα προμήθευσης και θα πρέπει οι νομοθετικές αρχές να το εξετάσουν αυτό. Η ρυθμιστική αρχή στην Ιρλανδία έχει την εξουσία και την ικανότητα να καθορίσει τις τιμές και κάθε αύξηση τιμής την εγκρίνει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Ιρλανδίας. Εγώ είμαι δραστήριος πολιτικά πάρα πολλά χρόνια. Πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκίνησα την πολιτική μου στα, σταδιοδρομία, ο υπουργό Ενέργειας στη χώρα μου καθόριζε ποια τιμή, σε ποια τιμή ε, θα αγοράζαμε την ενέργεια και ανταποκρινόταν αυτή η τιμή και στις συνθήκες της αγοράς και στις ανάγκες του καταναλωτή και όταν ήταν δύσκολα τα πράγματα έπεφταν οι τιμές. Ο καταναλωτής λοιπόν δεν έχει δει κανένα όφελος ακόμα από το υποτιθέμενο ανεξάρτητο ε, και ενιαίο ρυθμιστικό σύστημα, οργανισμό δηλαδή ρυθμιστικών αρχών. Ευχαριστώ κύριο Νίμπλερ παρακαλώ. Η κυρία Νίμπλερ με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για τις ενδιαφέρουσες, την ενδιαφέρουσα εισήγηση και τα ενδιαφέροντα σχόλια. Εμείς, ε, όπως ε, ίσως δεν ξέρετε, προέρχομαι από τη Γερμανία, έχουμε τη δική μας ενεργειακή πολιτική και με ενδιαφέρει η γνώμη σας. Πώς εκτιμάτε και από ρυθμιστικής απόψεως την αλλαγή της ενεργειακής ε, στρατηγικής στη Γερμανία ε, αποφασίσαμε να καταργήσουμε την ατομική ενέργεια και το 2022 θα έχουν πλέον σταματήσει τη λειτουργία του τα τελευταία εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ατομική ενέργεια ε, και είχαμε διαπιστώσει ότι έχουμε από τις ε, Εναλλακτικέ πηγές ενέργειας ένα πλεόνασμα το οποίο διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να το εξαγάγουμε στις γειτονικέ χώρες ε, και για οικονομικό όφελος, αλλά όταν παρουσιάζεται έλλειψη ε, ενέργειας σε ορισμένες περιφέρειες της Γερμανίας πρέπει να ξαναγοράσουμε αυτό το οποίο πουλήσαμε εμείς ως ε, ενέργεια σε ακριβότερη τιμή, μια εντρελοκομείο δηλαδή, το οποίο δεν είναι δομημένο, δεν είναι διαρθρημένο και δεν είναι σταθερό. Ε, όπως ίσως ξέρετε, υπογράφτηκε χτες ε, ο μεγάλος συνασπαλισμός ε, με την νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Και τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Η υπηρεσία αυτή, το ICER, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες χώρες, δηλαδή ασχολείται με έρευνες και μελέτες συγκεκριμένων χωρών όσον αφορά το ρεύμα, την παροχή, την επάρκεια ενέργειας δεδομένου ότι εδώ δημιουργούμε, φτιάχνουμε ορισμένα εμπόδια ώστε να διαφεύγει ρεύμα προς την Πολωνία, δηλαδή να, πηγαίνει, μην πηγαίνει χαμένο. Πρώτο ερώτημα λοιπόν, εάν επικεντρώνεστε, αν στοχεύετε σε συγκεκριμένες πολιτικές έναντι συγκεκριμένων κρατών και δεύτερον, θέλετε να εντατικοποιήσετε τη διασυνοριακή συνεργασία Δηλαδή, έχετε ασχοληθεί με το θέμα της ενίσχυσης ε, τη συνεργασία αυτή των ανταλλαγών ενέργειας, τη εμπορίας ενέργεια προς την Τσεχία. Ε, θέλετε να παράσχετε ε, καλύτερα κίνητρα για να ενισχυθεί αυτή η διακρατική, το διακρατικό παρεδόσε. Το υπερσυναριακό μάλλον παρεδόσε. Ευχαριστώ κύριε Σοντή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτές τις παρουσιάσεις. Καταλάβαμε λίγο το συσχετισμό μεταξύ καταναλωτού τιμής και του γεγονότος ότι δύσκολα μπορεί να περάσει σε άλλον προμηθευτή. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι συμβαίνει για το, με το συσχετισμό μεταξύ επενδύσεων και ρυθμισμένων τιμών. Πολύ συχνά διαβάζουμε στον τύπο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μια μέρα θα έχουμε μαύρη τρύπα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια μέρα θα έχουμε μαύρη τρύπα ενέργειας και ότι θα υπάρχει γενικό blackout γιατί οι προμηθευτές δεν θα έχουν πλέον πόρους. Τι σχέση βλέπετε να υπάρχει εσείς μεταξύ της, ε, των ρυθμισμένων τιμών, την ικανότητα επενδύσεων των ε, ιδιοκτητών υποδομών, δηλαδή λίγο πολύ των προμηθευτών, και τις ανάγκες να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις και καλύτερη διοργάνωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επίρου. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται και με τις σημερινές σχέσεις με την Gazprom προχωρεί στην ε, δημιουργία υποδομών και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένω. Τι γίνεται με τι υποδομέ και τι εγκαταστάσει σε ε, επίπεδο Ευρώπη. Διότι οι πολίτε, αλλά και εμεί οι βουλευτέ, κάποιε φορέ έχουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν αρκετέ επενδύσει. Παρά τι ε, αλλαγέ τη τάση κατανάλωση και παραγωγή. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Οντί. Ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις από πλευρά συναδέλφων. Θα ξαναδώσω το λόγο στους προσκεκλισμένους μας, στον κύριο Μόγκ, τον Λόρδο Μόγκ και τον κύριο Ποτόσνικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις διότι μεγάλο μέρος της εκθεσής μας ε, αφιερώνεται και σε αυτά τα θέματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Κάποιες ερωτήσεις νομίζω απευθύνονταν σε εμά. Βέβαια δεν μπορούμε να τι απαντήσουμε όλες. Απαντήσεις θα έπρεπε να έρθουν, κάποιες απαντήσεις θα έπρεπε να προέρθουν από άλλες ε, κατευθύνσει. Από την πλευρά του οργανισμού μας. Υπάρχουν, όπως είπα, δύο σημαντικά νομοθετήματα. Η τα οποία ήδη έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία υλοποίηση και υπάρχουν και δύο σημαντικότητα νομοθετήματα για την ηλεκτρική ενέργεια, για τις διασυνδέσει και την ε, διαχείριση της ε, κατανομής δυνατοτήτων. Αυτά θα περάσουν από την διαδικασία επιτροπολογίας πολύ σύντομα, το ίδιο και για το φυσικό αέριο, μια αντίστοιχη οδηγία. Όπως ξέρετε, έτσι κι αλλιώ δεν είναι στο χέρι μα να ελέγξουμε τι θα γίνει με τη διαδικασία τη επιτροπολογία στο φορέα μα για τι τιμέ του αερίου. Θα το σχολιάσω από διαφορετικέ σκοπιέ. Έχουμε παρατηρήσει μετακίνηση από τις παλιές ε, τιμές, τις συνδεδεμένε, σε τιμές αυτές που θα ονομάζαμε hub διότι η αγορά εδώ και μία χρονική περίοδο είχε μεγαλύτερες βραχυπρόθεσμες τιμές από ότι μακροπρόθεσμες τιμές που προέκυπταν από τις συμβάσεις. Καταλάβαιναν λοιπόν οι ίδιοι καταναλωτές όταν τους συνέφεραν οι τιμές hub, Στις περισσότερες από αυτού του είδους τις τιμές όμως δεν έχουμε την ευελιξία ώστε να γίνουν προφανές, ε, προφανές τιμές αναφοράς. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε από την πλευρά μας είναι αυτά τα hubs να χρησιμοποιηθούν, να είναι πιο ευέλικτα και και να διασυνδεθούν καλύτερα μεταξύ τους. Να είναι μια πιο ελκυστική αναφορά για τις ανάγκες της αγοράς. Τα διάφορα κενά που διαπιστώνουμε όμω στο σύστημα ε, δεν προκαλούνται μόνο από τα προβλήματα του ανέμου στην Γερμανία. Ε, εδώ χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση και, βραχυ, και μακροπρόθεσμη ταυτόχρονα. Η, η μόνη μόνιμη λύση όμως στο τέλος όλης αυτής της προσπάθειας θα είναι να έχουμε ευθύ δίκτυα. Προς τα εκεί οδηγούμαστε τόσο ή να συνδυαστούν οι δυνατότητες όλων των χωρών μεταξύ τους παράλληλα και θα το είδατε, αναφέρομαι στο γράφημα της σελίδας 15, δυναμικό, υπάρχει ακόμη και αφού έχει χρησιμοποιήσει ότι έχει να χρησιμοποιήσει η αγορά. Δηλαδή, πρέπει να συνδυάσουμε μεν τις διάφορες ε, ικανότητες που υπάρχουν, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Τώρα η αλλαγή, η μετατροπή, το πέρασμα σε άλλον προμηθευτή έχει να κάνει και με την συμπεριφορά των καταναλωτών, κάτι που είναι σχετικά ε, πρόβλεπτο. Έχουμε σημειώσει ποιε είναι οι τάσει ε, στην αγορά του αερίου. Έχω όμω εδώ να δώσω και δύο παραδείγματα. Εάν δείτε τη διαφάνεια 10 στο φάκελό σα, βλέπετε και φαίνεται περισσότερο στο αέριο αυτό βλέπετε ότι κοιτάξαμε αν υπάρχει σχετισμός μεταξύ των οικονομιών που μπορούν να κάνουν οι καταναλωτέ, περνώντα από τον ε, βασικό, από τον προμηθευτή στον οποίο βρίσκονταν αρχικά σε έναν φθηνότερο και στην Ευρώπη βλέπουμε να υπάρχει θετική αναλογία. Μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερε είναι οι οικονομίε που μπορούν να κάνουν οι καταναλωτέ, τόσο περισσότερο θα αλλάζουν προμηθευτέ. Υπάρχουν όμω κάποια στοιχεία που διαψεύδουν αυτή την τάση δεν θέλω να κατονομάσω καμία χώρα, αλλά κυρίω δεν μπορώ να αποφύγω παρά να μιλήσω για τη Γερμανία. Γιατί οι καταναλωτέ στη Γερμανία μπορούν να εξοικονομήσουν τόσο σημαντικά ποσά. Ε, το γνωρίζουν και δεν το κάνουν. Υπάρχουν και άλλες πτυχές λοιπόν. Η περιπλοκότητα της αλλαγή, το κόστος. Η ρύθμιση των τιμών παίζει κάποιο ρόλο, ακόμη και όταν δεν είναι ένα σοβαρό φραγμό με τη ρύθμιση των τιμών ο καταναλωτής έχει εμπιστοσύνη ότι πληρώνει τη σωστή τιμή. Οι ρυθμισμένες λοιπόν τιμές μπορεί να είναι φραγμός ως προς την είσοδο εφόσον το επίπεδο είναι τόσο υψηλό που γίνεται απαγορευτικό για την πρόσβαση στην αγορά αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι και ένα εστιακό σημείο ένα κομβικό σημείο και να δώσει μια ψευδέστηση εμπιστοσύνη και ασφάλεια στον καταναλωτή. Δεν πληρώνει περισσότερα από όσα θα έπρεπε να πληρώνει. Αυτό είναι το θλιβερό σκέλος της ιστορίας, ότι οι καταναλωτές δεν επωφελούνται από τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Αν όμως κανείς πάει παραπέρα, όχι απλώς επειδή έχουμε την έδρα μας στη Σλοβενία, αλλά αν δείτε το διάγραμμα 39, προς το τέλος του φακέλου, θα δείτε μια καθησυχαστική εικόνα για το τι συνέβη πέρυσι στην Σλοβενία. Ξεκίνησε μια νέα εταιρεία, προσέφερε στις τιμές του αερίου μια έκπτωση 20% και βασικά η αγορά ενώ βρισκόταν σε τέλμα ξαφνικά αναθερμάνθηκε. Και μέσα σε λίγες εβδομάδες 5% η, το ποσοστό της αλλαγής έφτασε το 5%. Πολύ καλό επίπεδο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μπορεί λοιπόν κανείς να ξεφύγει από το αδιέξοδο, να βγει από το τέλμα, εάν υπάρχει σωστό συνδυασμό ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, ρύθμιση και ανταγωνισμού. Σωστών ε, συνθήκων για να ευνοηθεί ο ανταγωνισμό. Η ιστότοπη με τι συγκρίσει των τιμών, α πούμε, είναι μια πολύ καλή επιλογή σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, στο ερώτημα εάν εμείς επικεντρώνουμε την πολιτική μας σε συγκεκριμένε χώρες. Βεβαίως, οι εθνικές πολιτικές αποτελούν τμήμα του μηχανισμού μας. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ρυθμιστικές αρχές όλων των 27 κρατών μελών, αλλά δεν είναι ο στόχος μας να εκδίδουμε ε, συστάσεις για μεμονωμένες χώρες εκτός εάν μας το ζητήσουν συγκεκριμένα. Ε, τέλος, αναφερόμενος στο θέμα των πόρων μας, στην αρχή του έτους ήρθα εδώ να παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασία μας και ξέφρασα τις ε, ανησυχίες μου επειδή δεν είχαμε επαρκείς πόρους να καλύψουμε τους στόχους μας, το έργο μας. Τώρα είμαι πολύ ικανοποιημένος να πω ότι με κάποιες καθυστερήσεις η Κομισιόν βρήκε τους αναγκαίους πόρους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την εντολή μας και πιστεύω ότι θα έχουμε αυτές τις πιστώσεις ε, ε, του χρόνου. Ε, λυπάμαι αν παρέλειψα κάτι, αλλά πιστεύω ότι απάντησα όσο μπορούσα. Ο, ο Λόρδος Μόγκ. Θα έπρεπε αντίθετα να ενεργήσουμε και να είχαμε ξεκινήσει με διαφορετική σειρά. Όσον αφορά εφαρμογή, ε, τότε βεβαίως η ελοποίηση υπάρχουν θέματα που προκύπτουν ιδίως προς τη λήξη της θητείας του Κοινοβουλίου και δεδομένου ότι εμπλέκεται και η Επιτροπή. Από πλευράς ρυθμιστικών αρχών εμείς δεν θα σταματήσουμε θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όσο το δυνατόν ταχύτερα και πιστεύω ότι και η Κομισιόν έχει καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για την ταχύτερη διεκπαιρέωση ε, της ε, υιοθέτηση και υλοποίησης των ε, προγραμμάτων, ιδίως προς αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Δεν θέλω να ξεκινήσω μια κριτική των θεσμικών οργάνων, πιστεύω όμως ότι ο τομέα τη υλοποίηση έχει βελτιωθεί. Ακόμα πολλά μπορούν να γίνουν. Όσον αφορά το switching, δηλαδή την αλλαγή του προμηθευτή στους καταναλωτές, εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε το υψηλότερο επίπεδο τέτοιων ενεργειών. Αλλά δεν είναι στρεβλωμένος ο ανταγωνισμός, διότι οι καταναλωτές, οι πολίτες που ήξεραν τα κόλπα και πώς να κάνουν την αλλαγή, το κάνουν πολύ συχνά, ενώ οι άλλοι δεν κάνουν καμία τέτοια αλλαγή, διότι είναι ανενημέρωτοι. Γι' αυτό θα πρέπει οι εταιρείε να υιοθετήσουν μια πιο δίκαιη πολιτική, να θέσουν στόχους καλύτερων επιδόσεων και ακόμα πιο σημαντικό και το λέω αυτό από πλευρά Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να κάνουν μία προσπάθεια να ανακτήσουν την ε, αξιοπιστία τους έναντι των καταναλωτών. Η... Το, συνεργ... το όραμα συνεργασίας, λυπάμαι που αναφέρω πάλι ένα όραμα, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα συνεργασίας ε, πρέπει να έχουμε πιο ξεκάθαρες θέσεις από την ε, πλευρά των προμηθευτών έναντι των καταναλωτών. Λυπάμαι που επανέρχομαι στις τιμές, στην τιμολόγηση, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάτω από το 50% των τιμών λιανικής πώληση, του κόστους δηλαδή της τιμολόγησης έχει σχέση με περιβαλλοντικό κόστος, κόστος δικτύου, κόστος ενέργειας, ε, ε, ε, πρωτοπαραγωγικών πηγών κλπ. Η ουσιαστική κίνηση που σημειώνεται στο 46% είναι στην χονδρική τιμή και αυτό είναι ο τομέας στον οποίο βλέπουμε τεράστιες ε, μετακινήσεις τιμών. Και όπως ε, ε, ελέγχθη από έναν συνάδελφο όσον αφορά τη, τη θέση του τομέα της βιομηχανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπουμε να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτρέπει μια πολύ βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά. Το επίπεδο των τιμών και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ξεπερνούν τις αρμοδιότητες και ικανότητες των μετριοπαθών ρυθμιστικών αρχών. Δυστυχώς. Και όσον αφορά τώρα την προστασία των καταναλωτών και ιδίως των ευάλωτων μερίδων του πληθυσμού, εδώ βέβαια λαμβάνονται διάφορα κοινωνικά μέτρα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να, εντοπίσουμε συγκεκριμένα πού είναι αυτοί οι ευάλωτοι πολίτες. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε συγκεκριμένους ε, πολίτες όταν δεν μπορούν να αντιποκριθούν στο ενεργειακό κόστος. Αυτό ε, σαφώς είναι στρατηγική της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων. Το Ενωμένο Βασίλειο και άλλες έξι χώρες έχουν ε, εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για να ερευνήσουν αυτά τα θέματα μέσω μιας ε, ιδιωτικής εταιρείας και δεν είναι σαφής ε, αυτές οι διακοιμάνσεις των αναγκών που υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και των έξι αυτών χωρών ε, συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό των προβλημάτων και των ανισοτήτων. Το τελευταίο σχόλιο που έχω αφορά τη γερμανική θέση. Οι κυβερνήσεις έχουν το απόλυτο δικαίωμα να αποφασίσουν ε, την πολιτική τους. Και αυτό που εμείς μπορούμε να μάθουμε από τις διάφορες ενέργειες είναι η ανάγκη της ολοκλήρωσης, της ενσωμάτωσης της ενεργειακής αγοράς. Βεβαίως ε, μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η θέση και η κατάσταση της γερμανικής αγοράς, το θέμα της εξάρτησης ε, από διάφορους πηγές ενέργειας αλλά η μία ολοκληρωμένη αγορά θα δημιουργηθεί μόνο όταν μπορέσουμε να ε, ομαλοποιήσουμε τους τρόπους λειτουργίας. Πριν από 10 χρόνια όταν έθεσα το ερώτημα της ενεργειακής ασφάλειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μου, υπέδειξαν διάφορα άθρα από τις εφημερίδες ε, από τα οποία θα μπορούσα να πληροφορηθώ του τι συμβαίνει. Τώρα έχουμε προχωρήσει σε ρυθμιστικό επίπεδο, σε ένα κανονιστικό πλαίσιο, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή επάρκεια. Εμείς ε, είμαστε ανεξάρτητοι ρυθμιστικοί φορείς και διαβουλευόμεθα με την Κομισιόν με καλή προδιάθεση βεβαίως για να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Έχουμε βεβαίως ξεφύγει από το χρονοδιαγραμμά μας, αλλά έχουμε την κυρία Τζόρνταν, η οποία θέλει οπωσδήποτε να κάνει μία ερώτηση και θα τη δεχτούμε. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα του κυρίου Τούρμες για τα κενά στη ροή, τα loop flows, διαφάνεια υπαριθμό 17. Εκεί λέτε την εξή δήλωση. Όταν αυξάνονται τα μη προγραμματισμένα κενά στη ροή, αυτό είναι κάτι που απαιτεί επίγουσες λύσεις και περισσότερη διαφάνεια. Και όταν σας ρώτησαν γι' αυτό, είπατε ότι δεν προκαλεί και ένα στη η αιωλική ενέργεια μόνο. Μας λέτε και τίποτα άλλο. Μπορείτε να εμβαθύνετε. Είναι τεχνικό το ζήτημα, το ξέρω. Αλλά ε, θα γίνουν δράσεις, θα αναλάβουν δράση οι θύνοντες, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων. Απάντηση ερευνούμε την πηγή των κενών στη ροή. Αυτά έχουν αυξηθεί σημαντικά στην κεντρική και στην ανατολική Ευρώπη, ειδικότερα στην Πολωνία, στην Σλοβακία, στη Δημοκρατία της Τσεχίας, στην Ουγγαρία, στην Αυστρία και προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις. Με αισθητήρε προσπαθούμε να μάθουμε γιατί υπάρχουν αυτά και από πού προέρχονται. Είναι φυσικό φαινόμενο, αν θέλετε, στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Αφύσικος είναι ο βαθμός στον οποίο έχει ενταθεί το φαινόμενο αυτό. Και απαιτεί σχεδόν το σύνολο της ε, χωρητικότητας που διατίθεται εκεί, ε, της εμπορικής. Και προσπαθούμε να έχουμε άμεση δράση, δηλαδή μια άμεση μετατροπή όταν υπάρχει κενό στην Πολωνία να ε, αλλάζει ε, η βάνα αν θέλετε και να μεταφέρεται αυτόματα το αντίστοιχο οι σοβαρές ενέργειες από τη Γερμανία και του Μπαλίν. Ε, προσπαθούμε δηλαδή να λύσουμε το πρόβλημα βραχυπρόθεσμα αλλά πρέπει να αρθούν τα τελικά ουσιαστικά τα εμπόδια για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς και θα πρέπει να βρούμε και ένα ε, τρόπο να αποζημιώσουμε αυτούς που πλήττονται από αυτά. Όσοι ζητούν ε, ε, αποκατάσταση πληρώνονται, αποζημιώνονται, αλλά δεν αλλάζει η πηγή της προέλευσης των κενών αυτών. Δηλαδή θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη αυτοί που δημιουργούν αυτά τα κενά και άρα μας χρειάζεται περισσότερη συνεργασία για να λυθεί το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση η τελική λύση θα πρέπει να είναι ένα πιο ισχυρό δίκτυο, ένα πιο ισχυρό σύστημα, έτσι ώστε οι ροές ενέργειας να μεταφέρονται χωρίς να φτάνει στο κόκκινο ε, το δυναμικό, το εθνικό ε, προμήθευσης ενέργεια, το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με αυτά τα κενά. Ωραία, ολοκληρώσαμε αυτό το πρώτο τμήμα της απογευματινής συνεδρίασης. Σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας και για την ε, προθυμία σας, κύριε Ποτότνε και Λόρδε Μόγκ. Και θα σας ξαναδούμε σε επόμενη ευκαιρία. Bene, iniziamo il nostro lavoro. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας από εκεί που είχαμε σταματήσει το πρωί για το Horizon 2020. Να ξεκινήσουμε με το Cesar. Έχουμε για τη συζήτηση αυτή στη διάθεσή μας 20 λεπτά. Να δώσουμε απευθεία το λόγο στη συνάδελφο Τόμσεν. Το σύστημα ΣΕΖΑΡ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Ενιαίας Κυκλοφορίας, είναι μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με στόχο να ε, βελτιωθεί η εναεριακή κυκλοφορία. Υπάρχουν ανεπάρκειες στον κατακαιρματισμένο ενιαίο χώρο της Ευρώπης και αυτό στοιχίζει 5 δις ευρώ ετησίως στις αεροπορικές εταιρείες και προστίθενται χιλιόμετρα στην απόσταση που διανύει μια μέση πτήση. Άρα και καίγονται περισσότερα καύσιμα, υπάρχουν μεγαλύτερες εκπομπές, ε, υπάρχουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις, πολλά, ε, πολλές δηλαδή παρελκόμενες επιπτώσεις. Ε, θα υπάρξει χάος στον χώρο τα, στα αεροδρόμια θα υπάρξει συμφόρηση, δύο εκατομμύρια πτήσει θα είναι αδύνατο να απογειωθούν ή να προσγειωθούν εάν συνεχιστούν τα πράγματα προ αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό πρέπει ο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο να γίνει πιο αποτελεσματικό. Χρειάζεται έρευνα για να υπάρξει απαραίτητη τεχνολογία, για να έχουμε έναν ευρωπαϊκό εναέριο χώρο πιο καθαρό, πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό. Οι πτήσει ε, πρέπει να είναι φθηνότερε και πιο ασφαλεί. Η έρευνα σε αυτό αποσκοπεί, επιτρέποντα για παράδειγμα στι αεροπορικέ εταιρείε να ε, ακολουθήσουν τη διαδρομή που επιθυμούν στην πτήση, την πιο άμεση, την πιο γρήγορη και στην έκθεσή μου δίνω έμφαση σε τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, ε, σύγκρουση συμφερόντων Δεύτερον, διασύνδεση με το πρόγραμμα για, ορίζοντα για το 2020. Και τρίτον, ε, σημασία που έχει η ενθάρρυνση πιο πράσινων τρόπων μεταφοράς. Ως προς το πρώτο, θα πρέπει να δηλωθεί η παρουσία ή η απουσία συγκρούσεων συμφερόντων από τον κάθε ενδιαφερόμενο που συμμετάσχει. Και θα πρέπει οι δηλώσεις ε, ε, συμφερόντων να κατατίθενται εκ των προτέρων θα πρέπει τα θέματα της ισότητας του φύλου να μπουν στην ημερήσια διάταξη και στα συμβουλευτικά όργανα και σε τα δικαιοδοτικά όλα. Το ίδιο ισχύει και για το ΣΕΣΑΡ. Θα πρέπει ε, βάσει του άρθρου 16 του ορίζοντα για το 2020 να ε, είμαστε σίγουροι ότι η διάσταση του φύλου θα ληφθεί σωστά υπόψη. Και βεβαίως οι προτεραιότητες για την καινοτομία της, του ορίζοντα, με ορίζοντα το 2020 δηλαδή πιο ε, έξυπνοι, πιο ολοκληρωμένοι, πιο πράσινοι τρόποι μεταφοράς. Ε, θα πρέπει αυτές οι αρχές και οι προτεραιότητες να εφαρμοστούν εδώ και στην ε, εναρία κυκλοφορία. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τόμψεν. Το λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Στοζινόφσκι, οπότε σας δίνω ευθύς αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Προφανώς το θέμα είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό, το πρόγραμμα CESAR και πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε να βασίζεται η, η βιομηχανία αερομεταφορών σε περισσότερα επιστημονικά δεδομένα που θα επιλύουν τα προβλήματα και τα θέματα. Απ' την άλλη πλευρά το ΣΥΖΑ ε, δημιουργήθηκε με το στόχο ότι το 2016 τα, οι επιστημονικοί στόχοι θα ε, συγκεραστούν, θα, θα δημοσιευθούν σε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και τώρα το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει ολοκληρωθεί και θα ήρθε ο καιρός να κάνουμε μια ενδελεχή ανάλυση για να δούμε σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα και τι είδους πρόοδο πρέπει να επιτύχουμε για τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ποιες άλλες επιστημονικές ε, ερευνητικές δραστηριότητες θέλουμε να ενισχύσουμε. Πρέπει να έχουμε ένα όραμα, ένα πρόγραμμα, ε, στόχους συγκεκριμένους για τα ερευνητικά προγράμματα ε, συμφωνώ και υποστηρίζω απολύτως όλα τα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί ή εγκριθεί μέχρι τώρα, αλλά παρόλα αυτά χρειαζόμαστε μια πολύ προσεκτική και ενδελεχή ανάλυση για τους στόχους μας και τη χρηματοδότηση στο μέλλον. Τώρα, η χρηματοδότηση προέρχεται από διάφορους ε, πόρους και γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε σαφώς τι θέλουμε να κάνουμε με αυτά τα κονδύλια. Και θα πρέπει το χρονοδιάγραμμα να ε, επεκταθεί, να διευρυνθεί και ως όδηση συγητής από τη δική μου πολιτική ομάδα υποστηρίζω την ουσία και θα προσπαθήσω να εδραιώσω τη διαφάνεια όσο τον δυνατόν καλύτερα και τώρα εκφράζω την υποστήριξή μου ε, στον εισηγητή και ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει η διαφάνεια όσο το δυνατόν πιο ισχυρή. Ισχυρό στοιχείο. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο του Σνόφσκι. Τώρα ο συνάδελφος Τζόρνταν. Ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω για τις δικές μου απόψεις, αλλά για τον κύριο Κάτσα. His views about this... Κάντσιο, από την ομάδα του ΕΛΚ. Εν όψη των τελευταίων εξελίξεων και δεδομένου στις αερομεταφορές έχει επιτευχθεί πάρα πολύ αργή πρόοδος και δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι κατά την άποψη του κυρίου Κάνσιαν. Ε, θέλουμε να επιτύχουμε επιτέλους αποτελέσματα. Ο κύριος Καντσιάν πιστεύει ότι η πολιτική βούληση δεν επαρκεί για την όλη ολοκλήρωση του μηχανισμού και γι' αυτό η συνέχιση αυτής της δομής και στη χρηματοδότηση και στους ανθρώπινους πόρους είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο κύριος Κάντσιαν επίσης πιστεύει ότι το ΣΕΖΑ, η κοινή επιχείρηση, έχει λειτουργήσει καλά, έχει παράσχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και γι' αυτό προτείνει την πρόταση της Κομισιόν να ανανεωθεί, να, να διευρυνθεί χωρίς καμία αλλαγή. Κατά την περίοδο του 2007-2012 η εμπειρία μας έδειξε ότι ο χρηματοδοτικός μηχανισμός μέσω των συμπράξεων ιδιωτικού δημοσίου τομέα ε, λειτουργεί και ότι στηρίζεται ε, σαφώς την υποβολή προτάσεων μέσα στο 7ο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Επίσης, ο κύριος Κανσιάν υποστηρίζει την ε, συνέχιση των προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και όσον αφορά τώρα τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς, βλέπουμε ότι δεν έχουν σημειωθεί τίποτα ανησυχίε ή επιφυλάξεις για την οικονομική διαχείριση του ΣΕΣΕΡ, άρα και εκεί δεν χρειάζονται αλλαγές, τροποποιήσεις. Ένας άλλος λόγος ε, υποστήριξη της ε, προτάσεως είναι ότι το πρόγραμμα ΣΕΖΑ θα αρχίσει πλέον τη φάση ε, υλοποίησης και ανάπτυξης και θα ήταν λάθο να επιτρέψουμε τυχόν νομοθετικά κενά ή εκκρεμότητε θα πρέπει, δεν θα πρέπει να διακυβεύσουμε με κανέναν τρόπο την προσεκτικά μελετημένη φάση ανάπτυξης του ΣΕΖΑΡ και γι' αυτό ο κύριος Κανσιάν είναι υπέρ της υιοθέτησης των προτάσεων της Κομισιόν χωρίς καμία τροποποίηση. Ευχαριστούμε, συνάδελφο Καρβάλιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την Μπρίτα Τόμψεν Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους για τη σημασία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, του Single European Sky και της κοινή επιχείρησης CESAR. Όχι μόνο γιατί έχει ευρωπαϊκή αξία, αλλά και για το όφελος που προσφέρει στο περιβάλλον και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει να σχολιάσω ότι αυτή η κοινή επιχειρήση, όπως και οι προηγούμενες, θα πρέπει να βασιστεί στις αρχές που έχουμε συμπεριλάβει στο Horizon 2020. Κάποιες από αυτές ήδη αναφέρθηκαν από την εισηγήτρια και τους προαλήσαντες συναδέλφους. Διαφάνεια, απλούστευση, σημασία της τεχνολογίας, αρχή ανοιχτού πνεύματος σε όλες τις πτυχές και η πολλαπλή χρηματοδότηση ε, εφόσον μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό στόχο από διαφορετικές πηγές εφόσον θα ε, κάνει κάποια διαφορά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα η όλη προσπάθεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρος, ας ακούσουμε τώρα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Τόμψεν, για την πολύ ωραία έκθεσή της. Το ΣΕΣΑΡ, όπως είπατε κάποια από εσά, είναι πραγματικά η τεχνολογική βάση για την πρωτοβουλία Single European Sky. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όχι μόνο από την άποψη της, του εξυγχρονισμού του όλου τομέα, από τεχνολογική σκοπιά, αλλά και προκειμένου να παρασχεθεί ευρωπαϊκή να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοπορία στον τομέα της διαχείρισης της εναρίας κυκλοφορίας. Εδώ καλωσορίζουμε την ε, δήλωση, την εισήγηση που ακούσαμε από την κυρία Τόμψεν και απλώς να σχολιάσω κάποιες από τις τροπολογίες που προτείνει η συγγετρία, μόνο να διευκρινίσω κάποια πράγματα δηλαδή, για την τροπολογία 8, όπου, όπου υπάρχει αναφορά μόνο για το Horizon 2020. Να λάβουμε υπόψη ότι εδώ αυτή η κοινή επιχείρηση ήδη προβλέπεται και στηρίζεται στο 2016 από το πρόγραμμα TNT με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Να είμαστε λοιπόν συνεπείς για την τροπολογία 12. Καταλαβαίνουμε τα κίνητρα της εισηγήτριας να προβλεφθεί αυτή η διάταξη για να υπάρξει μεγαλύτερη ισότητα των φύλων και να προωθηθεί αυτό. Δεν έχουμε αντίρρηση, όμως θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο, την θέση της Προεδρίας πάνω απ' όλα, έχει να κάνει και με τις λειτουργίες της Επιτροπής. Οπότε η γενική διεύθυνση μου είναι κάπως υπεύθυνη για την Προεδρία σε αυτές τις περιπτώσεις. Για τις τροπολογίες 13 και 14 τώρα, για τις συγκρούσεις συμφερόντων. Θα πρέπει να πούμε ότι εδώ το θέμα αυτό ανέκαθεν ήταν προτεραιότητα για την ε, κοινή αυτή επιχείρηση και τα πάντα έγιναν με βάση τα σχετικά άρθρα του εσωτερικού κανονισμού. Οπότε, εφόσον τους κανόνες αυτούς τους ετοίμασε η ε, το υπεύθυνο ελεγκτικό συνέδριο σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση και τον Eurocontrol υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί ώστε να υπάρχει προστασία για περιπτώσεις ε, σύγκρουση συμφερόντων ώστε να ξέρουμε πώς να τις διαχειριστούμε να τις αποφύγουμε και να απαντήσω και σε μια παρατήρηση που έγινε από κάποιον βουλευτή για το πώς αναλύονται τα προγράμματα. Έχουμε πολλά στοιχεία στα χέρια μας που δείχνουν τα αποτελέσματα και την ε, πρόοδο της κοινή αυτής επιχείρησης και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει μια δεύτερη αποτίμηση του όλου προγράμματος η οποία θα διατεθεί όμως δυστυχώς του χρόνου ε, στην καλύτερη περίπτωση το ακριβές πρόγραμμα εργασιών για τις επόμενες φάσεις, για το επόμενο διάστημα δηλαδή, είναι κάτι που είναι αντικείμενο διαβουλεύσεων αυτή τη στιγμή με τους ε, ενδιαφερομένους. Θα περατωθεί στο πρώτο εξάμενο της επόμενης χρονιάς και εκεί θα υπάρξει και ε, προκήρυξη διαγωνισμού ε, για, πρόσκληση ενδιαφέρον, για υποβολή, πρόσκληση, υποβολή ενδιαφέροντος. Θα φροντίσουμε λοιπόν, ε, μόλις έχουμε περισσότερα στοιχεία, να σας ενημερώσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Η Μπρίτα Τόμψεν. Ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες στις παρεμβάσεις Πιστεύω ότι γενικά συμφωνούμε στο πλαίσιο συμφωνώ με τον κύριο Τσαφνόφσκι ότι πρέπει να κάνουμε όντως μία ανάλυση όπως πρότεινε για να δούμε ε, τι είδους νέα ε, έργα, νέα προγράμματα πρέπει να αναπτυχθούν αλλά συμφωνώ και με την ε, συνάδελφο του κυρίου Κανσιάν που μίλησε εκ μέρους του ότι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε πολλές αλλαγές διότι τα πράγματα έχουν καλώς όπως τα πρότεινε η Κομισιόν. Από πλευρά ε, τώρα, τι πρέπει να σημειώσουμε στην ατζέντη μας, πρέπει να ακολουθήσουμε το άρθρο 16 και το άρθρο 16 δεν είναι ε, τόσο ε, εύκολο για μας να το εφαρμόσουμε γιατί από πλευρά της Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει το, τη διάσταση του φύλου να την εφαρμόσουμε όποτε χρειάζεται. Άρα λοιπόν κυρία Καρβάλιο πράγματι σύμφωνα με τις γραμμές του 2020, του ορίζοντα 2020 θα, θα ενσωματώσουμε όλες τις ψυχές που είναι απαραίτητες σύμφωνα ακριβώς με, τις, με τα άστρα. Ευχαριστούμε την συνάδελφο. Να θυμίσω ότι η ημερομηνία προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 4 Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Και τώρα να περάσουμε στο, στη συνέχεια του ορίζοντα 2020. Έχουμε ένα πακέτο θεμάτων εδώ, ένα σύνολο θεμάτων. Ο συνάδελφος Τούρμες δεν είναι εδώ όμω αυτή τη στιγμή. Θα δούμε το θέμα του μετά. Να ξεκινήσουμε με τη συνάδελφο Φόρντ. Έχουμε στη διάθεσή μας μία ώρα και πέντε λεπτά ω τις πεντέμιση. Θα φροντίσουμε να οργανωθούμε έτσι ώστε να προλάβουμε πέντε λεπτά λοιπόν ανά εισηγητή και εισηγητρία. Κυρία Φόρντ, Um, thank you very Ευχαριστώ. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα να λάβω περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κλινικών δοκιμών που σχετίζονται με το ΣΥΖΕΣ και την εργασία που έχει γίνει στο παρελθόν ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες ακριβώς όπου απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα. Επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτές οι τρομερές ασθένειες, οι μεταδοτικές, ε, κατευθύνονται και προς την Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικές ε, να αντιμετωπίσουμε τις ε, παγκόσμιες προκλήσεις. Μάλιστα, μόλις την περασμένη εβδομάδα συζητήθηκαν ε, μερικά μελλοντικά φάρμακα τα τα οποία θα βοηθήσουν την καταλέμηση της σηματίωσης. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τους καλύτερους ευρωπαϊκούς πόρους ε, για να καταπολεμήσουμε αυτές τις ασθένειες. Υποστηρίζω ε, τους βασικούς στόχους και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους, ε, τους συναδέλφους που με βοήθησαν ε, από, διακομματικά από όλες τις ομάδες και επίσης ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Καρβάλιο η οποία ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα και η οποία εργάστηκε μέσα στα πλαίσια των χωρών ΑΚΕ και έχει παρακολουθήσει το πώς έχει εξελιχθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Στην έκθεσή μου προβάλλω ορισμένες από τις σκέψεις μου και θα ήθελα τα σχόλιά σας, δεν ξέρω αν ακολουθώ τη σωστή κατεύθυνση. Παραδείγματο χάρη στο παράρτημα αναφέρω ορισμένους στόχους για τις κλινικές δοκιμές που τέθηκαν σε, σε, για διάφορες χώρες. Αυτό δεν είναι απαραίτητα πρωτογενής στόχος διό, και μου είπαν ε, άλλοι πιο έμπειροι από το παρελθόν ότι δοξιμε, δο, κλινικές δοκιμές μπορούν να, γίνουν μεν και να ας πούμε συμπληρώσουν κάποια στοιχεία ή κάποιο ερωτηματολόγιο ή ε, στατιστικές χωρίς ουσιαστικά να ωφελήσουν τον πλησισμό. Ε, γι' αυτό θα μελετήσουμε προσοχή τις τροπολογίες εκείνων που είναι πιο έμπειροι από μένα. Επίσης ε, πρέπει να συντονιστούμε και με άλλες, ε, άλλους αρμόδιους φορείς και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα για τις κλινικές δοκιμές. Ορισμένες λοιπόν από τις αλλαγές που προτείνω ε, στοχεύουν στην βελτίωση του συντονισμού με άλλους οργανισμούς, με άλλες αρχές. Αυτό δεν έχει γίνει τόσο πολύ υπό το πρώτο πρόγραμμα και πρέπει να το βελτιώσουμε. Προσπάθησα να, ε, διατηρήσω το πλαίσιο της περιγραφής των ασθενειών αυτών όσο το δυνατόν ευρύ ώστε να έχουμε μία ευελιξία στην περιγραφή και τον ορισμό του διαβήτη παραδείγματος χάρη και το, τις σχέσεις του και τις επιπτώσεις του με άλλες ασθένειες διότι Υπάρχουν ε, πολλές ασθένειες οι οποίες συνδέονται μέσω ε, επιπτώσεων συμπτωμάτων με άλλες ασθένειες είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, να εφαρμόσουμε πρόσθετα μέτρα διαφάνειας, όλα αυτά τα, τα δέχομαι ως ιδέες ευχαρίστως και στην ιστοσελίδα του Ορίζοντα 2020 υπάρχει μια, ένα link που παραπέμπει στην ενημέρωση αυτού του θέματος. Ορισμένοι εισηγητές σήμερα το προείπαν ότι αντί να υπάρχει προθεσμία μέχρι το 2024 να, να την ε, ε στο, να την καθορίσουμε στο 2020. Εάν αλλάξουμε την προθεσμία δεν σημαίνει αυτό ότι θα μειώσουμε τη χρηματοδότηση, θα αλλάξουν οι κατευθυντήριες γραμμές. Αλλά ενδέχεται να μην μπορούμε να ολοκληρώσουμε μέχρι το 2020 και να χρειάζεται η αρχική προθεσμία 2024. Γι' αυτό θέλω να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Αυξημένη συμμετοχή, ναι. Αριθμητική στόχη ε, δεν είμαι βέβαιη, διότι έχουμε έναν ευρύ κατάλογο ασθενειών που δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να το μειώσουμε, ε, τον κατάλογο αυτό ή να το περιορίσουμε. Σα περιμένω λοιπόν ε, με ανυπομονησία τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστούμε. Ε, την κυρία Φόρντ, το λόγο έχει η κυρία Καρβάλιο, παρακαλώ. Ή, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ο κύριος Χάμσταρτ. Και μετά η Ιζαμπέλα και μετά η κυρία Καραβάλιο. Παρακαλώ. This uh, uh, Το θέμα αυτό το οποίο έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διεξάγουν έρευνα είναι υπεύθυνες υπεύθυνε για το 70 με 75% όλων των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες όμως που διεξάγουν έρευνα, σε αυτές οφείλεται το 4% ε, των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς μόνο. Άρα είναι δύσκολη η κατάστασή τους, ε, βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Και οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο καπιταλισμός όπου το κράτος έχει τόσο ισχυρή θέση όπως είναι το, η περίπτωση της Γαλλίας όπου το σύστημα είναι μεγάλο και όπου το μεγάλο σύστημα είναι αυτό που διαμορφώνει το σύνολο της οικονομίας, αυτή είναι η περίπτωση της Γερμανίας, και ότι ο, ο καπιταλισμός όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι όμιλοι έχουν τόσο ισχυρή θέση, αυτό είναι το μοντέλο το αγγλοσαξονικό, <coughs> αλλά και το σύστημα της Βορείου Ιταλίας είναι κάτι που μας ενέπνευσε, όπως και τα προηγούμενα, διότι στη Βόρειο Ιταλία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις uh, uh, δημιουργούν δίκτυα μεταξύ τους και συνεργάζονται, δικτυώνονται και λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά, παράγουν καινοτομία. δυσδύουν ε, στα κενά της αγοράς και τα καλύπτουν. Το πρόβλημα που τίθεται λοιπόν είναι το εξής. Αυτά τα προγράμματα που στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη δεν είναι προγράμματα ενοποιημένα, είναι διάσπαρτα, είναι κατακαιρματισμένα το σύστημα θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό, περισσότερο αποτελεσματικό. Υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των διαφόρων δομών. Έχουμε το Eureka, το Ευρίκα, ένα διακυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 1995 και στο οποίο συμμετέχουν 14 ευρωπαϊκές χώρες και το Ισραήλ εκεί, αλλά και μη ευρωπαϊκές χώρες όπως ο Καναδάς και η Νότια Κορέα είναι συνδεδεμένα μέλη. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και το πρόγραμμα της Eurostat, το οποίο θέτει στο επίκεντρό του τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη. Και σε αυτό το πλαίσιο, 33 χώρες εμπλέκονται σε αυτό, το πρόγραμμα και εκτός από τις 33 χώρες μέλη του Ευρύκα ε, συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος, πλήρες μέλος και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χρηματοδότηση. Το πρώτο πρόγραμμα της Eurostat ξεκίνησε το 2008 και τώρα έχουμε ε, διανύουμε την τελευταία χρονιά της πρώτης προγραμματικής περίοδου του προγράμματος. Δηλαδή το 2013 είναι η τελευταία χρονιά της πρώτης φάσης και έτσι συνδυάζονται τα ωφέλη του Ευρύκα με την εμπειρία 25 ετών η οποία έχει συσσωρευτεί εμπειρία ε, με δραστηριότητες που έχουν αναρριφθεί ε, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Σε εθνικό επίπεδο πρέπει να πω τα εξής. Οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης ε, καλύφθηκαν με 300 εκατομμύρια ευρώ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, δόθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ. Άρα είναι πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε τις συμπράξεις, τη, μάλλον τη δημόσια με την ιδιωτική χρηματοδότηση ε, για να καλυφθούν ε, ακόμα και μικρότερες μονάδες. Με αυτά τα δημόσια κονδύλια. Πρέπει επίσης να πω ότι το πλαίσιο αυτό επεκτάθηκε διότι δόθηκε συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία με το Eurostat 2. Όλα τα ποσά τριπλασιάστηκαν που δόθηκαν σε αυτό το project. Άρα από την επόμενη χρονιά και μετά, από το 2014 μέχρι το 2020, Στο πρόγραμμα αυτό θα έρθουν κονδύλια σε εθνικό επίπεδο ύψους 860 εκατομμύριων ευρώ, 270 εκατομμύριων ευρώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα 1,1 1 δισεκατομμύριο 148 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο, το άθροισμα. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η πρόοδος. Και έτσι θα μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λογικά να υποφεληθούν από αυτές τις ε, δραστηριότητες. να υποφεληθούν από ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, αν θέλετε και ο οικονομικός αντίκτυπος είναι πολύ σημαντικός. Το πρόγραμμα της Eurostar θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ενίσχυση της εργασίας, της ανάπτυξη, της αηφόρου ανάπτυξης, στην ενίσχυση της απασχόλησης μάλλον και όλα αυτά ε, συνάδουν με τους στόχους της Ευρώπης για το 2020. Το Eurostars στην τελευταία ε, περίοδο 2008-2009 αξιοποίησε το Eurostar το πρόγραμμα αυτό 100 εκατομμύρια ευρώ δημόσια χρηματοδότηση και ιδιωτική χρηματοδότηση 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με ίδια κεφάλαια λοιπόν, ε, αναλήφθηκαν δράσεις. Στο Eurostar 2 Είχαμε δημόσια χρηματοδότηση από 33 συμμετέχοντα μέλη στο Ευρύκο, Ευρικά, στο, στο Ιουρίκα και όπως ανέφερα ήδη, 861 εκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο. Η πρόταση της Κομισιόν ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο φέτος και ε, απαιτούνται 270 ε, εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο λοιπόν 1,1 της περίπου και άρα βλέπετε ότι αυξάνεται σημαντικά η χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα αλλά και η ιδιωτική χρηματοδότηση η οποία συμμετέχει κατά 50% ε, στα επιλέξιμα κόστη των έργων. Και άρα και ο ιδιωτικό τομέα θα συμβάλλει με ένα ε, δισεκατομμύριο 148 εκατομμύρια ε, κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περίοδου, από το 2014 μέχρι το 2020. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία, οι βασικές πληροφορίες για το Eureka, για το Eurostar ε, και ως εισηγητής θα υποβάλω τρεις τροπολογίες. Πρώτον, άρθρο 5.2, ECE Top-Up και θα διαβάσω την τροπολογία, το κείμενο και παραθέτω. χωρίς να ξεπεράσει το, τη μέγιστη οροφή που ορίζεται στη παράγραφο υπαριθμών 1, κατά κανόνα η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ίση ή το 1 τρίτο της συμμετοχής των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7.1α και θα καλύπτει η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοικητικά και λειτουργικά κόστη τέτοιου είδου δαπάνες, και στην περίπτωση κατά, την οποία, ε, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος πρέπει να προσαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως μπορεί να διωθεί ευελιξία ε, κατά περίπτωση και θα μπορούσε κατά περίπτωση η συνεισφορά να φτάσει κατά μέγιστο στο ίμιση της συμμετοχής ε, των συμμετεχόντων κρατών, ενώ πριν θα είναι στο 1 τρίτο. Δεύτερη τροπολογία. Ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διεξάγουν έρευνα. Η πρόταση τη Κομισιόν στο άρθρο 2.2 είναι η εξή. Οι, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που διεξάγουν έρευνα είναι οι επιχειρήσει που θα επανεπενδύσουν τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών του ε, σε δράσει έρευνα και ανάπτυξη ή που αφιερώνουν ανα πάσα χρονική στιγμή 10% ε, του κύκλου εργασιών του σε δραστηριότητε έρευνα και ανάπτυξη. Η τροπολογία μου λοιπόν ως προς αυτό, ως προς την πρόταση της Κομισιόν, Δέκα λεπτά έχετε φτάσει, λέει η Πρόεδρος. Καλώς, τότε θα σταματήσω εδώ. Ε, μπορείτε να διαβάσετε την ε, τροπολογία μου, θα, θα τη δώσω γραπτός στα μέλη της Επιτροπής και θα έχετε την ευκαιρία να ε, είστε ενήμεροι. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και ελπίζω κάποιες προτάσεις και παρατηρήσεις να προκύψουν από αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον ε, συνάδελφο. Έχουμε κι άλλο λίγο χρόνο τελικά. Αλλά τώρα σε ακούσουμε την κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματος μετρολογίας και καινοτομίας είναι η παροχή λύσεων μετρολογίας που θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις καινοτομίες και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Υποστηρίζουν επίσης και τις τεχνολογίες μέτρησης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων όπως η υγεία, το περιβάλλον και η ενέργεια, όπου συμπεριλαμβάνεται η στήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή διαφόρων πολιτικών πρωτοβουλειών. Ένα σημαντικό στόχος της πρότασης είναι επίσης η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος έρευνας μετρολογίας σύμφωνα με το άρθρο 185 των συνθήκων με ενεργό συμμετοχή σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Μετρολογίας είναι ένα σημαντικό μέρος της δέσμης επενδύσεων καινοτομίας στο πλαίσιο του καινούριου προγράμματος πλαισίου Horizon 2020. Η αξιόπιστη και ανιχνεύσιμη μέτρηση επιτρέπει στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα να δημιουργήσει καλύτερα εργαλεία ούτως ώστε η επιστήμη και η έρευνα να καθίστανται πιο αποδοτικά. Αυτό το πρόγραμμα θα διαδεχθεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Μετρολογίας και θα συμβάλλει σε μια σειρά από εμβληματικές πρωτοβουλίες του πλαισίου Ευρώπη 2020 που επηρεάζονται από την έρευνα της μετρολογίας. Αυτό θα γίνει με την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, με την υποστήριξη της διαδικασίας τυποποίησης που δημιουργεί ευκαιρίες για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες. Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος θα διευρυνθεί περιλαμβάνοντας ενότητες αφιερωμένες στη βιομηχανική έρευνα και την εκμετάλλευση, στη στήριξη της τυποποίησης και στη δημιουργία ικανοτήτων. Επίσης, ο αριθμός των κρατών μελών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αυξηθεί από 22 σε 28. Όλες οι κυβερνήσεις σε τεχνολογικά προηγμένες χώρες υποστηρίζουν την υποδομή μετρολογίας λόγω των ωφελών που φέρνει ως δημόσιο αγαθό που δικαιολογεί τη δημόσια παρέμβαση. Μεγάλες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην έρευνα μετρολογίας και τις συναφείς υποδομές. Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των επενδύσεων στον τομέα αυτό και το ρόλο του στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας και της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, οι στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη-μέλη μονομερός. Η αριστεία που απαιτείται για την έρευνα και την ανάπτυξη λύσεων μετρολογίας εχμής έχει εξαπλωθεί πέρα από τα εθνικά σύνορα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. Χωρίς μια συνεπή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ψηλός κίνδυνος επανάληψης προσπαθειών με συνέπεια την αύξηση κόστους. Η προστιθέμενη αξία της δημόσιας παρέμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έγκυται στην ικανότητα να συγκεντρώσει στεγανά εθνικά ερευνητικά προγράμματα, να βοηθήσει στο σχεδιασμό κοινών στρατηγικών έρευνας και χρηματοδότησης πέραν των εθνικών συνόρων, και στην επίτευξη κρίσιμης μάζας των φορέων και των επενδύσεων που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ερευνητικά συστήματα μετρολογίας. Ταυτόχρονα στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών. Σημειώνεται ότι η Ένωση αναμένεται να συνεισφέρει το 50% της συνολικής χρηματοδότησης. Όσον αφορά το περιεχόμενο του σχεδίου έκθεσης, εξέτασα την πρόταση της Επιτροπής, εντόπισα ορισμένα τεχνικά ζητήματα για τα οποία έχω προτείνει ορισμένες τροπολογίες. Κυρίως, ο στόχος των τροπολογιών είναι να ευθυγραμμιστεί η πρόταση της Επιτροπής για τη Μετρολογία με αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί στις εκθέσεις του ορίζοντα 2020 που περάσαμε την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε την κυρία Τζαβέλα. Και τώρα η συνάδελφος Καρβάλιου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για το θέμα αυτό και ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, την κυρία Φόρντ συγκεκριμένα για το δεύτερο πρόγραμμα σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χώρων για τις κλινικές Δικημέ. Να πω ότι συμφωνώ πλήρως με όσα η κυρία Φόρντ έχει προτείνει, τα έχουμε συζητήσει και πραγματικά οι απόψεις μας εμπίπτουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε αυτό το, στην επεξεργασία αυτού του προγράμματος και όπως είπε και η κυρία Φόρντ, ευθύς εξ αρχής από το 2003 όταν ήμουν υπεύθυνη έρευνα στην Πορτογαλία έπρεπε να ασχοληθώ με τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του προγράμματος. Το γνωρίζω πολύ καλά, ξέρω ότι δεν πάει καλά και τι πηγαίνει καλά. Οπότε Θέλω να διευκολύνω όσο μπορώ με τις γνώσεις μου να βοηθήσω να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Είχα το προνόμιο πρόσφατα με την ε, Επίτροπο Γιώργαν Κουίν να επισκεφθώ περιοχές στην Αφρική όπου το πρόγραμμα αυτό ήδη υλοποιείται και πραγματικά εντυπωσιάστηκα με το έργο Ευρωπαίων ερευνητών και επιστημόνων σε πολύ δύσκολες συνθήκες πολλές φορές, αλλά πραγματικά προσφέρουν ε, υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους που τη χρειάζονται. Σε πολλές φορές σε παραγκουπόλεις γύρω από το Cape Town συγκεκριμένα, στην Νότια Αφρική, και πραγματικά ήταν συγκινητικό, διότι οι επιστήμονές μας που δημοσιεύουν άρθρα στο Nature και στο Science και καταφέρνουν να φροντίζουν ανθρώπους σε συνθήκες πολύ δυσχερείς πολλές φορές. Είναι λοιπόν μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω στην επεξεργασία αυτού του προγράμματος. Τι δεν πηγαίνει καλά τώρα, είναι αρκετά περίπλοκο. Στα πρώτα στάδια μας είχε πάρει μια τριετία για να ξεκινήσει το πρόγραμμα να λειτουργεί βάσει των ε, χρυσών ε, κανόνων που είχαμε θέσει. Από διοικητικής πλευράς είναι πολύ περίπλοκο και θέλαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απλουστεύσουμε, να υπάρχει λιγότερος διοικητικός φόρτος, γραφειοκρατικό άχθος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους συμμετέχοντες. Ξέρω ότι η απλούστευση είναι κάτι που επιδιώκεται και μετά το Horizon 2020, αλλά όταν ε, μπλέκονται κράτη-μέλη και ο ιδιωτικός φορέας πρέπει τα πράγματα να είναι απλούστατα για να λειτουργήσουν ε, σωστά. Η διαφάνεια και το ανοιχτό πνεύμα ήδη αναφέρθηκαν, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη που θα πρέπει να βελτιώσουμε. Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ραπτεξικό Ταμείο. Αυτό το ταμείο ε, χρηματοδοτεί πολλά θέματα υγείας και κλινικής, ε, κλινικών δοκιμών στην Αφρική. Όμως πρέπει να γίνουν εδώ κοινέ προσπάθειες. Διότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορεί να κάνει το ε, ευρωπαϊκό το πρόγραμμα για την σύμπραξη Ευρωπαϊκών για Αναπτυσσόμενων Χωρών, αλλά μπορεί να τα κάνει το Αναπτυξιακό Ταμείο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση το πρόγραμμα έχει πολλές, ε, πολλά σκέλη οικοδόμησης ε, δυνατοτήτων σε συνδυασμό με τα εθνικά προγράμματα. Δηλαδή μπορεί να έρθει να συμπληρώσει τα εθνικά προγράμματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν είμαι βέβαια αν δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και λίγη περισσότερη στόχευση, καλύτερη στόχευση. Αν δείτε τι γίνεται από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, λόγω χάρη τα πρόσφατα εμβόλια από το Glass Smith Klein για την ελονοσία. Αυτά ε, πέτυχαν γιατί ήταν πολύ καλά στοχευμένα. Το πρόγραμμα αυτό είναι περισσότερο πρόγραμμα συνάρθρωσης διαφορετικών πραγμάτων που συμβαίνουν ταυτόχρονα, αλλά δεν έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Ίσως να μπορούσαμε ε, να πάρουμε τις προσπάθειες των 100 μελών και να ε, κάνουμε καλύτερη στόχευση στο πρόγραμμα. Να παραμείνει ανοιχτό στις νόσους και παθήσεις, αλλά κυρίως αυτές που πλήττουν ενδεχομένως ε, ήδη την Ευρώπη, όπως ο Δάγκιος. Ε, γιατί σε κάποιες ε, ευρωπαϊκές περιφέρειες απαντάτε η νόσος αυτή. Εδώ λοιπόν πρέπει να δοθεί κάποια προσοχή και σε αυτό το σκέλος. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με όσα υπόθηκαν από τη δίκη για τη διάδοση και την διεύρυνση της συμμετοχής, τη διαφάνεια. Όμως, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα που αφορά και το Ευρωπαϊκό Αναπτύξιακο Ταμείο και κυρίως είναι θέμα απλούστευσης. Ίσως με καλύτερη στόχευση θα πετυχαίναμε πολύ περισσότερα. Αυτά τα τρία σημεία θα ήθελα να συνεχίσω να συζητώ με την εισηγήτρια στις συναντήσεις των σκιωθών εισηγητών. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Μαντουρέλ. Μαντουρέλ. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση της κυρίας Φόρντ. Να σας πω ότι η πολιτική μου ομάδα στηρίζει τη δουλειά της εισηγήτριας και να σας πω ότι συμφωνούμε απολύτως με τους προβληματισμούς της, με τις ιδέες της, αλλά και με την τοποθέτηση της κυρίας Καρβάλιο. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να προσθέσω μόνο ένα σχόλιο σε αυτά των συναδέλφων με τα οποία όπως σας είπα συμφωνώ απολύτως και το σχόλιο μου είναι το εξής. Εάν στην περίπτωση την οποία συζητήσαμε σήμερα το πρωί για την πρωτοβουλία για τα νέα καινοτόμα φάρμακα, το ΛΥΜΕ, εάν θεωρούμε ότι το δημόσιο συμφέρον θα πρέπει να είναι ο γνώμονας για όλα τα πράγματα που χρηματοδοτούμε, τότε στο πρόγραμμα συνεργασίας της Ευρώπης και των αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές, προβάλλεται το επιχείρημα εάν θα πρέπει να ενθαρρυνθεί αυτό το πρόγραμμα να υποστηριχθεί ακόμα περισσότερο. Είπε και η κυρία Καρβάλιο και η κυρία Φόρτ ότι μιλούμε για χρηματοδότηση για ασθένειες που κατά κύριο λόγο πλήττουν τις πιο ευπαθείς ε, κοινωνικές ομάδες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και γι' αυτό θέλω να τονίσω το εξής. Η προσπάθεια αυτή έχει νόημα μόνο άμα τελικά θα υπάρξει πρόσβαση στα φαρμακευτικά προϊόντα και στις ιατρικές υπηρεσίες γιατί να μας χρησιμεύει ένα νέο εμβόλιο για την φυματίωση, για να αναφέρω την ίδια νόσο που ανέφερε και η κυρία Φόρντ, εάν το εμβόλιο αυτό συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό βάρος για μια οικογένεια, η οποία τελικά δεν μπορεί και να τα αγοράσει και άρα δεν μπορεί να της γίνει και το εμβόλιο αυτό για να προστατευθεί. Ε, πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει ο κανονισμός να το διευκρινίσει και από αυτή την έννοια λέω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα υποβάλουμε τροπολογίες. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που μας είπε ο κύριο Ράνσντορφ και το πρόγραμμα του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις δυνατότητες διεξαγωγής έρευνας. Καταρχάς η Eurostat θα βοηθήσει στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και υπηρεσιών στην αγορά. Όταν το συζητήσαμε, είπαμε ότι χρειάζεται να κοιτάξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διαφορετικό, υποδιαφορετικό φως, είτε μιλούμε για το, το πρόγραμμα ορίζοντας 2020, είτε όχι. Ε, δεν επαρκεί μια πολιτική δήλωση που να λέει ότι ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικές, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των μικρομεσαίων και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να επιβιώσουν από μια στρατηγική που θα ξεκινάει από τη βάση, από τις ε, ρίζες. Να διευκολύνουμε λοιπόν τις διαδικασίες για να εξασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Δεδομένου ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δεν έχουν νομικά, ένα νομικό τμήμα ή τις απαραίτητες υποδομές για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες. Ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, εξειδικευμένο δηλαδή σε όλες τις πτυχές αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να εξετάσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζει αυτό το πρόγραμμα και να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν πρακτικά. Θα επανέλθω με, έναν, με διάφορες τροπολογίες, με ένα αριθμό τροπολογιών προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μακοβίτσου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συζητητές για αυτά τα οποία είπαν. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, επειδή είμαι σκιώδης συζητητής στο πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την έρευνα. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω ε, σαφώς αυτό το κοινό πρόγραμμα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα όταν έχουμε πάρα πολλά άτομα χωρίς ε, δουλειά και ε, χωρίς ελπίδα ε, για το μέλλον να τις ενισχύσουμε. Και το πρόγραμμα της Program has been tailor-made for innovative SME. Και το πρόγραμμα STAR έχει βοηθήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε πολλές ε, συζητήσεις ε, εδώ στο Κοινοβούλιο για τις μικρομεσαίες και είμαι ευτυχής να πω ότι αυτό το πρόγραμμα Eurostar έχει επιτύχει συγκεκριμένα ε, αποτελέσματα και ελπίζω να συνεχιστεί και να παρουσιάσει ακόμα περισσότερα καλά αποτελέσματα. Στο πρώτο πρόγραμμα Eurostars, Eurostars 3,5 εκατομμύρια, 3.500 αιτήσει είχαν υποβληθεί και 800 αιτήσει, 800 υποβολές ε, προτάσεων χρηματοδοτήθηκαν ε, οι οποίες βασικά ήταν ε, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλες ήταν ερευνητικά Ινστιτούτα και φορείς. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε από τη βάση προς τα πάνω, ιεραρχικά δηλαδή. Δεν υπάρχει... Ε, δεν υπάρχει η προτεραιότητα για την χρηματοδότηση πρέπει να βαστίζεται στην ποιοτική αξιολόγηση. Τώρα το Eurostars 2 θα έχει ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι τρεις φορές μεγαλύτερος και έτσι θα δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν οι πιο καινοτομικέ επιχειρήσεις σε, αυτό, ε, σε αυτή την περίοδο κρίσης. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν και τις επιπτώσεις της κρίσης, ιδιαίτερα στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Πρέπει να γνωρίζουμε, να αναγνωρίζουμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να επιβάλλουν μεγαλύτερες περικοπές από, άλλες, από άλλα κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει αυτές να υπονομεύσουν τα αποτελέσματα του Eurostars 2. Επίσης ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλές φορές υπάρχει μία επικάλυψη αρμοδιοτήτων όταν έχουμε ε, ειδικέ και επιπλέον συμμετοχές από κράτη-μέλη. Οπότε υπάρχει μία σύγχυση για το ποιος ε, έχει την αρμοδιότητα να πράξει τι. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε έναν σωστό έλεγχο χωρίς κενά και ο εισηγητής προτείνει επίσης μία αύξηση στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διοικητικό κόστος. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη επίσης να κάνουν μία διάμεση αξιολόγηση. Οι ευθύνες τις οποίες θα αναλάβουν οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα Eurostar, Eurostars έχει δείξει ε, ε, ότι θα πρέπει, έχει αποδείξει σαφώς την αξία των ε, καινοτομιών και ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γκλάν. Γκλάντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Σαβέλα για το πρόγραμμα ΕΜΠΗ. Θα ήθελα να τονίσω την σημασία αυτού του προγράμματος, α, την κυρία Τζαβέλα, συγγνώμη, την κυρία Τζαβέλα, για το πρόγραμμα μετρολογίας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η ανάπτυξη αυτού του προγράμματος, διότι οι ακριβείς μετρήσεις είναι πολύ σημαντικές για να δώσουν το έναυσμα δραστηριοτήτων σε πολλές επιχειρήσεις. Ε, ε, επίσης την δανοτεχνολογία η αποθήκευση δεδομένων και εκεί παίζει σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό ακριβώς είδαμε πως αξιολογήθηκε ε, το πρόγραμμα που είχαμε μέχρι τώρα. 117 προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν από το 2009-2012 και πάρα πολλά ερευνητικά Ινστιτούτα έλαβαν μέρος σε αυτά τα προγράμματα, 22 ε, κρατών μελών. Η πρόταση της Κομισιόν για την συνέχιση του προγράμματος αυτού την ε, θεωρώ πολύ ικανοποιητική και δεν νομίζω να χρειάζονται μεγάλες τροποποιήσεις στην πρόταση της Κομισιόν. Δεδομένου ότι μόλις συμφωνήθηκε όλο αυτό το πακέτο ορίζοντας 2020, θέλω να πω ότι εδώ έχουμε συμφωνήσει συγκεκριμένους κανόνες για την έρευνα που μπορούμε να εφαρμόσουμε και στη μετρολογία. Ε, για τα άρθρα 185 και 187 επί των οποίων συζητούμε σήμερα, ε, πρέπει να διαπιστώσουμε πού είναι η κόκκινη γραμμή και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην την ξεπεράσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω το Eurostars πρόγραμμα σε συνδυασμό με το Ευρύκα Ευρικά είναι λίγαν αξιόλογο και χαίρομαι ιδιαίτερα που περισσότερα κράτη-μέλη συμμετέχουν σήμερα. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως θα πρέπει να διευρυνθεί, να επεκταθεί και στα μέλη του Eureka ή Εύρικα, έτσι ώστε να έχει και μια ε, διεθνή διάσταση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που διεξάγουν έρευνα. Πιστεύω ότι αυτό θα παρουσιάσει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το δικαίωμα τη διοικητική διαχείριση. Ήδη το πρωί μιλήσαμε για αυτά, τα πλεονεκτήματα αυτά, παραδείγματο χάρη στα ΣΔΙΤ, στι συμπράξει δημοσίων ιδιωτικών τομέων. Μπορούμε να κάνουμε μια μεταφορά κονδυλίων ε, ώστε να εφαρμόσουμε μια ευθυγραμμισμένη γραμμή χρηματοδότηση. Βέβαια το θέμα είναι πόσε υποβολές προτάσεων θα έχουμε στα πλαίσια αυτά των GTIs τα μεγάλα προγράμματα κατά κάποιο τρόπο θα αξιολογηθούν διαφορετικά από τα μικρά. Το θέμα είναι να έχουμε πολλές προτάσεις και όσον αφορά το 25 ή 33% της δημόσιας ενίσχυσης, αν μπορεί να δοθεί ή όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, ποια θα είναι η συμμετοχή του δημοσίου. Ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εμείνουμε στον άκαμπτο ορισμό του 10% ε, δεδομένου ότι το κόστος της έρευνας και οι δαπάνες της έρευνας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι σε μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό πρέπει να εισαγάγουμε το παράγοντα ευελιξία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες και δαπάνες. Γενικά νομίζω ότι το πρόγραμμα Eurostars είναι ενδεδειγμένο, αποτελεσματικό, γρήγορο και θα λειτουργήσει θαυμάσια. Όπως η πρώτη φάση, έτσι και η δεύτερη. Παραδείγματο χάρη, μειώνονται συνέχεια οι προθεσμίες πληρωμής, καταβολής δηλαδή των κονδυλίων. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά θετικό στοιχείο. Ευχαριστούμε κυρία Τόγια. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ. Ε, θέλω οπωσδήποτε να πω ότι χρειάζεται εξέταση της πρότασης που μας έγινε, διότι πρέπει να αξιολογηθούν οι συσχετισμοί που έγιναν και με τα ενδιάμεσα στάδια ε, στο επίπεδο του Eurostar 1 και από την πλευρά των εμπειρογνωμόνων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δείχνει, ε, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το πρόγραμμα ενδέχεται μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και στο Eurostar 2 κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό, ε, βοηθά και εξυπηρετεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι ένα διασυνοριακό δίκτυο το οποίο μπορεί να επιτρέψει την κοινοτομία μέσω της έρευνας. Είναι λοιπόν νομίζω σημαντικό η δεύτερη αυτή φάση του Eurostar που τώρα ξεκινά να ε, στηριχθεί σωστά. Όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι, θα πρέπει να επιδιώξουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση και καλύτερη συνάρτηση των διαφορετικών προγραμμάτων μεταξύ τους, ώστε να έχουμε περισσότερη υποστηθέμενη αξία. Αυτό θα συμβεί μόνον εάν πραγματικά δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα υπερκρατικό. Ε, και είναι νομίζω σημαντικό να διευρυνθεί το πρόγραμμα και να συμπεριλάβει και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε κάτι που με τις τροπολογίες μας θα επιδιώξουμε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς θα υπάρξει το ε, αποτέλεσμα αυτό μόχλευσης ως προς τη χρηματοδότηση που είχε το Eurostar 1. Θέλουμε αυτό να συνεχιστεί, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλό είναι να συμμετέχουν στα δίκτυα της έρευνας μεν, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, αλλά εφόσον υπάρξουν ήδη ερευνητικές διαδικασίες και εντοπιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, θα, μετά πρέπει να δούμε και πώς θα βρεθεί χρηματοδότηση, ιδίως από το δημόσιο φορέα. Γιατί ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι κυρίως οι επενδύσεις και το που θα βρει κανείς επενδυτικούς πόρους για να προχωρήσει. Και μετά θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ως προτεραιότητα την απλούστευση. Κάτι που το λέμε πάρα πολύ εδώ στην Ευρώπη, αλλά σπανίως το υλοποιούμε επαρκώς. Απλούστευση λοιπόν για να προσπαθήσουμε να, έχουμε, να αποφύγουμε διπλούς ελέγχους, επιβαρύνσεις που δεν χρειάζονται χρειάζονται σε τίποτε. Ε, και επίσης διασφαλίσεις ότι τα πράγματα πάνε καλά. Διότι όσο πιο πολύ περιπλέκονται οι κανόνες, όσο πιο πολύ ε, ε, πολλαπλασιάζονται τα επίπεδα ελέγχου, τόσο περισσότερο αυξάνονται και πιθανότητες επικάλυψης. Κάτι που δεν έχει κανένα νόημα. Απλούστευση λοιπόν και προσοχή στο διοικητικό κόστος. Νομίζω ότι το θέμα του διοικητικού κόστου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Αφορά ολόκληρη την έρευνα και όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί κάποιε φορέ το διοικητικό κόστος φαίνεται να είναι... Ε, σχετικό με την ποσότητα, ενώ πολλές φορές δεν έχει σχέση με τις διαστάσεις του δικτύου. Εδώ απαιτείται λοιπόν πολύ διαφάνεια, πολύ αυστηρότητα και πολύ μεγάλη προσπάθεια μείωση ε, του, διοικητικού, του κόστου. Εάν δεν κάνει το οργανόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σελίδε επί σελίδων με ονόματα προσωπικού, αν ρωτήσετε κανεί τι γίνεται με αυτή τη διοικητική μηχανή που είναι τόσο πολύ επιζήμια κατά την άποψή μου. αυτά είναι τα θέματα που ήθελα να γύρω. μετά από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και να επαναλάβω όλε αυτέ οι κοινέ επιχειρήσει, οι ενισχυμένε κοινέ επιχειρήσει θα μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην όλη προσπάθεια τη κοινοτομία για να μείνουν ε, ορθέ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δείξουμε και εμείς ότι πραγματικά κάτι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, την οικονομική κρίση στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφος Έλερ. Ähm, Πολύ σύντομα θα ήθελα να συμπρόσω και εγώ μετά την παρέμβαση του συναδέλφου Γκλάντε, Γκλάντε εκ μέρους του ΕΛΚ και στη συζήτηση με τους συντονιστές ε, θέλω να σημειώσετε ότι όλα αυτά τα θέματα τα βλέπουμε ως πακέτο, πακέτο. Δεν είναι μόνο απόφαση των εισηγητών, αλλά είναι και μια συμφωνία την οποία εμείς τουλάχιστον έχουμε με τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και πιστεύω ότι και με τις άλλες πολιτικές ομάδες συμμερίζονται αυτή την άποψη. Θέλουμε μία κοινή διαδικασία, δεν θέλουμε τα GTI και τα PPP να τα διαχωρίσουμε, τα Z δηλαδή, αλλά να τα διασυνδέσουμε όλα μαζί με τις κοινέ επιχειρήσεις um <coughs> ως πακέτο ενσωματωμένο με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και να μπορέσουμε να το διευθετήσουμε μέχρι τον Απρίλιο. Αυτό θέλω να τονιστεί και ε, ε, να σημειωθεί επίσης και από τους εκπροσώπους Κομισιόν και του Συμβουλίου. Η θεώρησή μας ως πακέτο. Ο κύριος Τούρμες, ε, μερικά σχόλια για τη δική του έκθεση που είναι εισηγητής. Ε, ευχαριστώ. Συγγνώμη που άργησα λιγάκι, αλλά είχα μία προθεσμία, είχα μία συνάντηση την οποία δεν μπόρεσα να αλλάξω και γι' αυτό είχα παρακαλέσει να συζητηθεί το θέμα μου για την ε, ανάπτυξη ενεργού και υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης λίγο αργότερα. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι αυτή είναι μία πρόθεσή μας ε, να ένα στόχος μας να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερα αυτά που γίνονται μέχρι τώρα. Σε αυτό τον τομέα έχω συζητήσει και με οργανισμούς και ε, αρχές οι οποίες ασχολούνται με ηλικιωμένους ανθρώπους και προσπαθούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση μεταξύ του να μπορέσουμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ή ευάλωτο άνθρωπο να τον κρατήσουμε στο σπίτι του ε, με την παροχή όλων των μέσων τεχνικής βοήθειας τα οποία χρειάζεται για να μπορέσει να ζήσει και να μπορέσουμε να εντάξουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους μέσα σε μία δομή μαζί με άλλους συνομήλικους. Μου λένε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ρίσκο, ένα ρίσκο να οδηγήσει η τεχνολογία σε μια παρακολουθούμενη μοναξιά. Δηλαδή μια μοναξιά του ατόμου η οποία θα παρακολουθεί τη συνέχεια με κάμερες ας πούμε ή με, τεχνητά, με τεχνολογία, με τεχνολογικά μέσα ώστε να παραμένουν οι ηλικιωμένοι ακόμα μεγαλύτερο διάστημα ε, στο σπίτι τους και θα παρακολουθούνται από μακριά δεν ξέρω αυτή, αν αυτός είναι ένας πραγματικός κίνδυνος, αλλά θέλω να το συζητήσω με τους άλλους συζητητές. Η τεχνολογία την οποία αναπτύσσουμε πρέπει πάντοτε να λαμβάνει υπόψη πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τους ηλικιωμένους μέσα σε μια κοινότητα, ε, μέσα σε, μια, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και να χρησιμοποιηθεί μεν η τεχνολογία όπως το Skype ας πούμε στο σπίτι για ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν αλλά μην απομονώσουμε κοινωνικά τους ηλικιωμένους λόγω προηγμένης τεχνολογίας. Το δεύτερο ζήτημα ε, πάντοτε όταν εμπλέκεται η τεχνολογία και η υποβοηθούμενη διαβίωση είναι σε ποιον ανήκουν όλα αυτά τα δεδομένα βάσει των οποίων θα κρίνουμε παραδείγματο χάρη το στοιχείο της ιδιωτικότητας είχα πει στη συζήτηση ότι τα δεδομένα αυτά ανήκουν στους ε, πελάτες οι οποίοι είναι οι πολίτες. Δεδομένου ότι αυξάνεται η φτώχεια στην Ευρώπη, αυξάνεται το κόστος ενέργειας, γίνονται συζητήσεις τώρα στην Ευρώπη αν όλη αυτή η τεχνολογία που υποτίθεται ότι διατίθεται για να διευκολύνει τη ζωή των ηλικιωμένων οδηγεί πάλι σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Είναι ενεργοβόρα δηλαδή. Γι' αυτό θέλω να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε φορά που αναπτύσσεται νέα τεχνολογία να μην ξεχνιούνται αυτές οι πτυχές της ε, ε των ενεργειακών πόρων. Εν συνεχεία, το θεσμικό πλαίσιο Τι θα γίνει αν ένα κράτος μέλος δεν συμμετάσχει σε αυτό το πολύ καινοτομικό πρόγραμμα ε, ή ε, υπάρχουν επιχειρήσεις ας πούμε που είναι top στην καινοτομίε και δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτά τα προγράμματα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να βρούμε μία λύση να μην αποκλειστεί κανένα ερευνητικό κέντρο ή Ινστιτούτο Καινοτομιών σε ένα κράτος μέλος που δεν θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή που η κυβέρνηση δεν θέλει. Χρειάζεται λοιπόν μία λύση ώστε να μην αποκλείσουμε κανένα φορέα που ενδιαφέρεται για να συμμετάσχει. Ε, εγώ βεβαίως ε, προσπαθώ πάντοτε να, να προβάλλω τα προβλήματα για να μπορέσω να δημιουργήσω κάποια δράση και αντίδραση. Σύμφωνο με τον κύριο Έιλερ ότι ως κοινοβούλιο θέλουμε να προωθήσουμε αυτό το ε, θέμα της συμμετοχής στο, στα πρόγραμμα αυτά για αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους ε, συμμετοχή δηλαδή στην έρευνα και στην ε, ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων, διότι είναι ευάλωτες μερίδες πληθυσμού που πρέπει οπωσδήποτε να βοηθηθούν. Ο συνάδελφος Μπερτζίνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα που αφορά πολλά κράτη-μέλη ταυτόχρονα. Ένα κοινό πρόγραμμα. Δυστυχώς το δικό μου κράτος δεν συμμετέχει. Παρόλο που όπως και ο κύριος Τούρμες θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα σημαντικότατο. Παρόλα αυτά θέλω να εκφράσω την ε, γνωσύνη μου για όσα έχει κάνει ο εισηγητής και έχω και μία παρατήρηση. Διότι σε κάποια σημείο οι απόψεις μας διαφέρουν με αυτές του εισηγητή. Το πρόγραμμα παρεκκλίνει από τους κανόνες του Horizon 2020 και υπερισχύουν οι εθνικοί κανόνες. Γι' αυτό το λόγο πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκουν το πρόγραμμα αυτό ελκυστικό. Εάν αλλάξει αυτή η διάσταση του προγράμματος, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι θα είναι αρνητικές οι συνέπειες. Ίσως λοιπόν ο εισηγητής μας θα μπορούσε να το ξανασκεφτεί. Έχει νόημα αυτό που προτείνει, διότι μπορεί να υπάρξει η ιδεατή συμμόρφωση με τους κανόνες, αλλά όχι το αποτέλεσμα που επιδιώκαμε τελικά. Επίσης, πιστεύω ότι ο εισηγητής προτείνοντας λύσεις για τα άριστα ιδρύματα των κρατών που δεν είναι μέλη του προγράμματος, που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό γιατί χρειάζεται και δημοσιονομική γραμμή και κάποιο υπεύθυνο ε, ως σύνδεσμος μεταξύ του δικτύου και των ιδρυμάτων. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος έλλερ πάλι. Δεν θέλω να συμπληρώσω αυτά που είπε ο συνάδελφος, αλλά να τονίσω ότι ο συνάδελφος υπέβαλε μια εξαιρετική έκθεση και ιδίως το θέμα της προστασίας δεδομένων, data protection, πρέπει να το προσέξουμε, διότι τα ιατρικά στοιχεία για ηλικιωμένους ανθρώπους πρέπει να τύχουν προστασίας ε, ε, και εγγύσεων. Είναι ευαίσθητα στοιχεία. Τώρα, η τηλεμετρική, η τηλεμετρική παρακολούθηση του, της καρδιάς, παραδείγματο χάρη, και η εξαποστάσεως καταγραφή των δεδομένων αυτών είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία δεν πρέπει να πέσουν σε λάθος χέρια. Αυτή η τηλεμετρική ιατρική λοιπόν είναι ένα σημαντικό στοιχείο και πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα στοιχεία. Είναι στοιχεία τα οποία είναι εξαιρετικά ιδιωτικά, δηλαδή εμπίπτουν στην πιο ιδιωτική σφαίρα της ζωής ενός ανθρώπου και γι' αυτό θα πρέπει να ίσως προωθήσουμε ειδικά μέτρα προστασίας των ιδιωτικών στοιχείων αυτών και της προστασίας των δεδομένων. Διότι ενδεχομένως ορισμένοι ε, ορισμένες από αυτές τις ομάδες των ηλικιωμένων δεν μπορούν μόνοι τους να προστατεύσουν, δεν έχουν ούτε την εμπειρία ούτε τις δυνατότητες να προστατεύσουν τα δεδομένα τους. Γι' αυτό θα πρέπει πάντοτε να κοιτάξουμε το θέμα της προστασίας δεδομένων όταν θέλουμε κοινωνικά να γίνουν αποδεκτά αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστούμε. Και τώρα λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Μετή για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τα γενικότερα σχόλια που διατύπωσα σήμερα το πρωί για το άρθρο 187, να έχουμε όλοι μας υπόψη την ανάγκη απλούστευσης, να καταβάλουμε όλοι προσπάθειες για να μάθουμε από την πρώτη γενιά, αν θέλετε, της εφαρμογής του άρθρου 185 και να φτάσουμε σε ένα κοινό μοντέλο όλο και περισσότερης εναρμόνισης μεταξύ όλων αυτών των πρωτοβουλειών και να αποφύγουμε τις αλληλοεπικαλύψεις με, τα, ε, την κείμενη νομοθεσία. Ορισμένες γενικές παρατηρήσεις πρώτα και μετά ε, πιο σχετικές για την κάθε μία από τις πρωτοβουλίες. Ως προς το άρθρο 185, δύο σημεία. Πρώτον, η ex έλεγχη. Η κατασταλτική δηλαδή έλεγχη. Ο οικονομικός κανονισμός επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει ασφάλεια στην, σε επενδύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιου είδους εγχειρήματα. Επομένως, η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει ε, ελέγχου και επαλήθευσης. Άρα, πρέπει να επανεξετάσουμε την ακαιρεότητα των ε, συστημάτων ελέγχου ε, της διαχείρισης των κονδυλίων και να διενεργούμε προληπτικούς ελέγχους εξάντε και ενίοτε και κατασταλτικούς εξπόστ. και δεν θα πρέπει να υπάρχει η αρχή της αιρεσιμότητας σε σχέση με τους ελέγχους ε, για την αξιοποίηση των κονδυλίων. Δεύτερον, το Ταμείο Εγγυήσεων είναι σημαντικό Όμως, βάσει του άρθρου 185 δεν μιλούμε για ευρωπαϊκούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Υπάρχουν όμως ε, κάποιες ε, επικίνδυνες, θα έλεγα, περιπτώσεις, όπως είναι το EDCP, και εκεί ο οικονομικός κανονισμός περιγράφει εναλλακτικέ λύσεις. Σε εθνική βάση, δηλαδή, μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα. Μπορούμε να βρούμε κάποια μέσα να το ρυθμίσουμε σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για το EDCP, ε, την έκθεση του κύριου Φόρντ, την οποία καλωσορίζουμε. Δύο λόγια. Ως προς τους στόχους, ε, μπήκε και ένα ερωτηματικό εδώ. Εάν θυμάστε την έκθεση του πρώην βουλευτή κυρίου Φαν υπήρχε μια διάμεση αξιολόγηση του EDCP1 και εκεί τόνισε ο πρώην βουλευτής ε, την έλλειψη των στόχων. Και γι' αυτό εμείς ως Κομισιόν βάλαμε τους στόχους για να αποκαταστήσουμε αυτό το παλαιότερο η κυρία Καρβάλιο μας μίλησε για την ανάγκη περισσότερης ε, συνέργειας και συνεργασίας με το Ταμείο ε, για την ε, ανάπτυξη την περιφερειακή και συμφωνούμε απολύτως. Τώρα για το Eurostar 2 έχει συζητηθεί πολύ εκτεταμένα. Συμφωνούμε με την άποψη του εισηγητή, το πνεύμα του, τη φιλοδοξία του. και υπάρχει δεσμεύση ε, τα συμμετέχοντα μέλη πράγματι να ε, ε, συμμετάσχουν, να, υπάρχουμε, να πάμε σε μια ενοποίηση, σε μια ολοκλήρωση, όχι συνεργασία, ένα βήμα παραπέρα. Βέβαια, ως προς τον προϋπολογισμό θα προτιμούσαμε τη διατύπωση του Eurostar 1 ως προς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 25% για να αυξηθεί ε, το ε, μοχλευτικό αποτέλεσμα έναντι των κρατών μελών. Τώρα ως προς την εθνική συμμετοχή. Ε, καλό θα είναι να ξεκαθαρίσουμε την ορολογία που χρησιμοποιούμε. Στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020, συνδεδεμένες χώρες είναι ε, μία λέξη που χρησιμοποιούμε με πολύ συγκεκριμένο νόημα, θα το θυμάται σίγουρα ο κύριος Χαλέρ, και δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τις συνδεδεμένες χώρες με κάποιες χώρες που συνδέονται με το Eureka, είναι μέλη του Eureka αλλά δεν είναι συνδεδεμένες χώρες βάσει του ορίζοντα 2020. Να πούμε λοιπόν ότι είναι χώρες ε, συνέτεροι, χώρες εταίροι. Ε, εταίροι κυρίως και από εκεί και πέρα, το bottom upness, από κάτω προς τα πάνω. Ο κύριος ε, Γιώχανσον το τόνισε αυτό. Το Eurostar δεν επιλέγει το θέμα, είναι βασικό χαρακτηριστικό, δεν επιλέγει το μέγεθος, είναι πολύ φιλικό προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές μπορούν να διαλέξουν σε ποιο χώρο θέλουν να διεξάγουν την έρευνά τους και αυτό είναι το βασικό ε, διαφοροποιητικό στοιχείο. Και τέλος, ο εισηγητής προτείνει μια λίστα ελέγχου ε, του κατά πόσο ε, πληρούνται ορισμένα κριτήρια, checklist και να δούμε αν μπορούν να ενσωματωθούν αυτές οι δυνατότητες. Αλλά αυτό έχει ήδη προβλεφθεί στο 2020 και στους στόχους του ορίζονται για το 2020. Άρα είναι μια επανάληψη χωρίς ε, πολύ νόημα κατά τη γνώμη μου. Έρχομαι τώρα στην έκθεση του κυρίου Τούρμες. Τρία σύντομα σχόλια. Χαιρόμαστε διότι το κείμενο ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για την Καινοτομία και αυτό είναι πολύ καλό. Στηρίζουμε ακραδάντως το κάλεσμα του κυρίου Τούρμες οι χρήστες να εμπλακούν ακόμα περισσότερο και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το, αυτό που χαρακτηρίζει τον κύριο Τούρμες και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και δεύτερον, αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Μπρεζίνα, Υπάρχει κάποια αντίφαση. Θέλουμε παρέκκληση από το EL2. Θέλουμε την εφαρμογή των εθνικών κανόνων συμμετοχής για να υπάρξει ευρωπαϊκή στήριξη. Στόχος μας ήταν να είναι φιλικό προς το χρήστη αυτό το περιβάλλον, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνήθως δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα πλαίσιο και τώρα θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή την πρωτοβουλία, την οποία συνήθως δεν είχαν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό αυτό το πληρώνουμε με το τίμημα του να έχουμε προβλέψει μια παρέκκληση σε σχέση με τους γενικούς κανόνες. Αλλά είναι ένα τίμημα που αξίζει να πληρώσουμε. Τώρα, η ΕΑΛ είναι απολύτως ανοιχτή και στις άλλες χώρες. Αλλά δεν είναι δυνατό να υπάρξουν ευρωπαϊκά κονδύλια ε, σε κοινά προγράμματα τα οποία να κατευθυνόνται σε χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη, γιατί δεν υπάρχει εθνική και στρατηγική μονάδα με την οποία να υπογραφεί η Σύμβαση Ανάθεσης, η οποία θα οργανώσει και θα διαχειριστεί το πράγμα αυτό. Ε, προβλέπονται όλα αυτά στο 185. Η ολοκλήρωση είναι ένα εγχείρημα που ε, Καλή για συμμετοχή διάφορα κράτη-μέλη και μετά ε, φτάνουμε σιγά σιγά προς τα πάνω. Αλλά σαφέστατα τα κράτη-μέλη πρέπει να το υπογράψουν. Δηλαδή μας δεσμεύει αυτός ο κανόνας. Όπως είπα σήμερα το πρωί, οι συνάδελφοι και εγώ είμαστε διαθέσιμοι οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση και να ευχαριστήσουμε θερμά όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου για τη συμβολή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μέτιου. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να ξαναδώσουμε το λόγο στους εισηγητές μας. Η συνάδελφος Καβάλη θέλει να δευτερολογήσει, παρακαλώ. Ναι, έχω μια ερώτηση προς την κυρία Ford, για την έκθεση μάλλον της κυρίας Φόρντ. Ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας βοηθήσει με μια πρόταση για το πώς να, το Ταμείο ε, Εγγύησης θα μπορούσε να ε, ισχύσει εδώ. Ανησυχούμε πολύ για το EDCP και εάν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ε, διαθέσιμες εγγυήσεις μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, διευκολύνει με τις τροπολογίες που θα υποβάλουμε ώστε να ξέρουμε πώς θα μπορέσει να αξιοποιηθεί. Μάλιστα. Μισό λεπτάκι, κυριολεκτικά μισό λεπτάκι, αν θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ναι, ναι. Ε, θα το συζητήσουμε με την κυρία Φόρτ και με σας κυρία Καρβάλιου. Υπάρχει τεχνική δυνατότητα. Ανέφερα τα εθνικά ε, προγράμματα και το δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίο και αυτό έχει κάποιε διατάξει σχετικά ε, και θα το πετύχουμε, πιστεύω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Όταν βρείτε απάντηση σε αυτό αυτήν την ερώτηση και κάποια λύση στο θέμα. Παρακαλούμε να μας, να μας ενημερώσετε και εμάς μεσογραμματίας. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Φόρ νομίζω έφυγε από την αίθουσα. Λάντσφορντ, Ζαβέλα και Τούρμες. Ο κύριος Ράσφορντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω πολλές παρατηρήσεις. Ε, τις κατέγραψα όσες προέκυψαν από τη συζήτηση. Για τη διαδικασία αυτή είναι ένα δημοσιονομικό εργαλείο αυτό μας δίνει ε, ένα, ε, ε, ένα μείγμα συμμετοχής και απόστασης στην ιστορία της επιστήμης και της ανάπτυξης ανέκαθεν το πρώτο πρόβλημα ήταν ο εντοπισμός του τομέα που έπρεπε να δράσει ένα ίδρυμα το θεσμικό πλαίσιο εδώ μπορούμε να ξεφύγουμε από το αυστηρά θεσμικό πλαίσιο και είμαι ευγνώμων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ετοίμασε αυτό το εργαλείο και μπορεί να αξιοποιηθεί. Δεύτερη παρατήρηση. Μια από τις τροπολογίες μου στόχο έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των εξαιρετικά μικρών επιχειρήσεων. Κάποιες επιχειρήσεις έχουν λιγότερους από 10 εργαζομένους Οπότε, ο κανόνας του 10% θα είναι πολύ δύσκολο να ε, ισχύσει στην περίπτωσή τους. Η τροπολογία μου λοιπόν αυτή ελπίζω ότι θα δώσει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Επίσης ελπίζω οι συνάδελφοι να στηρίξουν τη συγκεκριμένη λύση. Τρίτη παρατήρηση. Να θυμίσω ότι δεν πρέπει να ασκηθεί πίεση. Πίεση για την βελτίωση των εταιρικών σχέσεων, των κοινών επιχειρήσεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Είναι αδυναμία αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συγκρίνουμε το τι συμβαίνει εδώ και τι συμβαίνει στι ΗΠΑ λόγω χάρη. Ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι διαφορέ. Τέταρτη παρατήρηση. Ε, Ζωτική σημασία είναι να βγούμε από τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα αυτό και να συνεργαστούμε με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και τη Ρωσία βεβαίως. Ενημερώνομαι ότι ξεκίνησαν συνομιλίες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στον τομέα αυτό και οι Ρώσοι είναι φοβερά ε, περίεργοι να δουν τι μπορεί να γίνει με αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα με αυτό το ερευνητικό πλαίσιο μάλλον. Πέμπτη παρατήρηση. Αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια τη συζήτηση ήδη και το πρότεινα, πρότεινα διεύρυνση του πλαισίου ώστε να αντιμετωπιστεί το διοικητικό κόστος. Η διεύρυνση όμως του πλαισίου σκοπό δεν έχει μόνο το διοικητικό κόστος, αλλά τα ε, τέλη συμμετοχής. Δηλαδή, στο πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα συνδυασμένων προσπαθειών από διαφορετικές χώρες. Συμμετοχή λοιπόν διασυνοριακά. επιμέρους χωρών. Οπότε, ένα τέτοιο μέτρο σκοπό έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της συμμετοχής και των τελών συμμετοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον ε, συνάδελφο Ράνσπορτ για αυτή τη διεξοδική απάντηση και η κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι. Έλαβα υπόψη μου τα σχόλια των συναδέλφων και μαζί θα δουλέψουμε για το τελικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τούρμες. Θέλετε να απαντήσετε. Θα κρατήσω το χρόνο μου για μια επόμενη συζήτηση. Ωραία. Οπότε ολοκληρώσαμε επιτυχώς και αγκαίρως. Να ενημερώσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι το μεσημέρι στις 4 Δεκεμβρίου. Εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου. Επίσης η Επιτροπή Ήτρε θα συνέλθει αύριο στην αίθουσα 5G3 στις 9 το πρωί. 5G3 για να μην έχετε άγχος συνάδελφε.